Colleghi, ehm, possiamo cominciare il pomeriggio in... Ε, ξεκινήσουμε, έχουμε ένα έντονο και πολύ ενδιαφέρον απόγευμα. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του απογεύματο είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Εγκεμέν Μπαγκή, τον ε, Τούρκο Υπουργό για Ευρωπαϊκέ Υποθέσει και επικεφαλή ε, των διαπραγματεύσεων. Έχουμε και τον νέο πρέσβη που πρόσφατα διορίστηκε, τον κύριο Σελίμ Γενεράλπ, τον καλωσορίζω. Και φυσικά καλωσορίζω θερμά τον Υπουργό. Χαίρομαι που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας σε μια χρονική στιγμή όπου η Τουρκία ε, αποτελεί ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε την έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα σας, η Τουρκία, ε, στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Ο Όμεν Ρούιτεν είναι υπεύθυνος, υπεύθυ, υπεύθυνη για την έκθεση, τη χαιρετίζω. Κύριε Υπουργέ, στην, στο ψήφισμα του κυρίου Αλμπερτίνη που υιοθετήσαμε την περασμένη εβδομάδα, η Τουρκία αναφέρεται μαζί με τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες και έχει βασικά, βασικό, βασική θέση στο κείμενό μας και το μήνυμα που στέλνουμε είναι ένα μήνυμα ενθάρρυνσης για τα θετικά βήματα που έχει ήδη ολοκληρώσει σε διάφορα μέτωπα η Τουρκία και της δίνουμε ελπίζω και κάποια κίνητρα για να προχωρήσει σε περαιτέρω αλλαγές, ειδικά στον τομέα των, του δικαίου και των μειονοτήτων και τις θρησκευτικέ μειονότητες, την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την ελευθερία της έκφρασης και πολλούς άλλους τομείς. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να καλωσορίσω το ΕΚ Γιάν Όρμε, το συνάδελφο που είναι, της ε, Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων ε, του Ολλανδικού Κοινοβουλίου και Αντιπρόεδρο της, συνέλευσης του ΝΑΤΟ. Εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει στη συζήτησή μας, δεν τον βλέπω, αλλά τον καλωσορίζω παρόλα αυτά. Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Σας δίνω λοιπόν πάρα αυτά το λόγο και σας καλωσορίζω ακόμα μια φορά. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής, Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα και για τον νέο μας πρέσβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρισκόμαστε εδώ σήμερα, ειδικά μετά την θέση ενισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και τον ορισμό της δεύτερης Επιτροπής Μπαρόσο για να μιλήσουμε για ένα συναρπαστικό θέμα, την ένταξη της, Ευρωπαϊκή, της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Αλβερδίνη και τον κύριο Προβέρα, τον πρόεδρο και τον πρόεδρο της Επιτροπής μας φιλοξενούν εδώ πέρα σήμερα. Νομίζω είναι επίκαιρη η συνάντηση αυτή. Θα μοιραστούμε τα αισθήματα που έχουμε ο ένας για τον άλλον άμεσα. Εκτιμώ τις ε, συναντήσεις αυτές γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας ειδικά παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους λαούς Ευρώπης, από τους Ευρωπαίους πολίτες και η Επιτροπή σας έχει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης μας, νομίζω πως έχουμε πολλά να ε, συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για αλληλοκατανόηση, για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του λαού της Τουρκίας και οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις, ο διάλογος μεταξύ ημών και ημών θα παίξει κρίσιμο ρόλο στο να διασφαλίσουμε την αντίληψη μεταξύ των λαών μας και την αλληλοκατανόηση Πρόσφατα η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν εντείνει τις ε, σχέσεις τους και έχουμε άρα ένα βήμα καλύτερης κατανόησης, καλύτερης κατανόησης της Τουρκίας και της ένταξης της Τουρκίας και των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα. Επίσης η Τουρκία συζητιέται συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ανέφερε ο κύριος Προβέρα, Γι' αυτό πρέπει και εμείς να εκφράσουμε θέση μας σαφώς και ειλικρινά. Θα ήθελα και εγώ λοιπόν να ευχαριστήσω και την καλή μου φίλη, την κυρία Ρία Ομενρόιτεν, την εισηγήτρια για την Τουρκία που εργάζεται στο πολύ συναρπαστικό και ενδιαφέρον αυτό θέμα τα τελευταία χρόνια και έχει συνεισφέρει πολύ στην ενίσχυση αυτής της αλληλοκατανόησης. Αξιότιμα μέλη. Καθώς ξεκινάει η περίοδος της Λισαβόνας φαίνεται πως οι προτεραιότητες ή οι προκλήσεις της Ευρώπης είναι πως η Ευρώπη πρέπει να παίξει έναν παγκόσμιο ρόλο. Ε, υπάρχει ανάγκη για νέους δρόμους και πηγές ενέργειας, χρειαζόμαστε ασφαλή παροχή ενέργειας, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που μας απασχολεί όλους, η οικονομική κρίση και η ανάγκη για νέες αγορές, η ανεργία η λάθρομετανάστευση και η ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών στην Ευρώπη είναι σημαντικό θέμα. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι προσπάθειες καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην Ευρώπη. Η προώθηση της δημοκρατίας και της ορθής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου είναι όλα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Αυτές είναι οι κοινέ μας προκλήσεις και όταν σκεφτόμαστε αυτά τα προβλήματα η Τουρκία εμφανίζεται ως ε, ένα λαμπερό αστέρι γιατί είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ακόμη και πριν ενταχθούμε είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε σε όλους αυτούς τους τομείς και άλλους. Καθώς η συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, καθιστά την Ευρώπη ένα παγκόσμιο παίκτη, η Τουρκία έχει το πλεονέκτημα να είναι η μόνη χώρα που είναι ταυτόχρονα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, του ΟΣΑ, των G20, του Οργανισμού της Ισλαμικής Διάσκεψης και πολλών άλλων οργανισμών. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η Τουρκία είναι ακόμη και παρατηρητής στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών. Οπότε είναι πολύ ενεργοί. Είμαστε υπερήφανοι για τις διαμεσολαβητικές μας ειρηνευτικές προσπάθειες. Είχαμε τέσσερις γύρους συνομιλιών πρόσφατα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Μεσολαβήσαμε επίση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν και η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα που μπορούσε να φέρει αυτούς τους δύο ηγέτες στο ίδιο τραπέζι. Έχουμε αναλάβει για τρίτη φορά τη διοίκηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Διαπραγματευόμαστε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, Ρωσίας και Γεωργίας, Συρίας και Ιράκ, Βοσνίας και Σερβίας ταυτόχρονα. Ακόμα προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και το διάλογο μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν και του δυτικού κόσμου γενικότερα. Ο στόχος μας είναι λοιπόν ο ίδιος. Ίσως κάποιες φορές να έχουμε διαφορετικό ύφος λόγω των διαφορετικών παραδόσεων της δικής μας περιοχής του κόσμου που καμιά φορά μας δίνουν διαφορετικές έννοιες και αντιλήψεις, αλλά οπωσδήποτε η Τουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων εκεί πέρα. Όπως λέμε και στα τουρκικά, άμα καίγεται το σπίτι του διπλανού, κάτι πρέπει να κάνεις γιατί θα κάνει και το δικό σου. Προσπαθούμε λοιπόν να σβήσουμε τις φωτιές στην περιοχή μας. Η... Η παρέμβαση της Τουρκίας σε αυτή την περιοχή δεν υποκινείται από ιδεολογία, θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο, απλά από τα αμοιβαία συμφέροντα και την ανάγκη για ειρήνη. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο ειρηνικό έργο της ανθρωπότητας. Εάν αναλύσετε γιατί ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί είναι τόσο επιτυχημένη μέχρι στιγμής είναι γιατί απέτρεψε τον περαιτέρω πόλεμο σε αυτή την Ήπειρο. Και σε αυτό πιστεύει και η Τουρκία. Η Τουρκία πιστεύει πως μπορούμε και εμείς να αποτελέσουμε μέλος της ομάδας μαζί σας για την ειρήνη και για την πρόληψη μελλοντικών πολέμων. Είμαι σίγουρος πως όσοι από ε, σας παρακολουθείτε την συζήτηση περί της Τουρκίας είστε περίεργοι και για την Κύπρο. Όπως ε, ξέρετε το κόμμα του οποίου είμαι μέλος έχει την εξουσία από το 2002. Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία κάναμε όταν αναλάβαμε την εξουσία ήταν να προσαρμόσουμε την στρατηγική μας όσον αφορά το Κυπριακό. Υποστηρίξαμε τις ε, προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα να προετοιμάσει το σχέδιο Ανάν, τους ενθαρρύναμε να ξεκινήσει και τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των μερών, που οδήγησε στην προετοιμασία του σχεδίου Ανάν. Ενθαρρύναμε τους τουρκοκυπρίους να ψηφίσουν υπέρ του σχεδίου Ανάν και μετά την αποτυχία αυτού του σχεδίου, λόγω της απόρριψης του από τους Ελληνοκύπριους φίλους μας, ακόμα ενθαρρύναμε την ε, ηγεσία του Βορρά να συνεχίσει συνομιλίε. Και οι πρόεδροι Ταλάτ και Χριστόφια έχουν συναντηθεί 50 φορέ πέρσι μόνο, το τελευταίο έτο. Και υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε λοιπόν μια συνολική λύση στο νησί το συντομότερο δυνατόν. Αλλά αυτό πρέπει να βασίζεται στην δικαιοσύνη. Η κοινή έκκληση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να βρεθεί μια λύση με βάση μια διζωνική, δικοινοτική μια τέτοια λύση είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε με πολιτική ισότητα. Θέλουμε λοιπόν ο πρόεδρος Ταλάτ και ο ομόλογος του να καταλήξουν σε μια λύση που θα σέβεται τις κοινότητές τους και η Τουρκία θα υποστηρίξει την επιλογή των Κυπρίων. Βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή των συνομιλιών αυτών και προσωπικά είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω πω οι δύο θαραλέοι αυτοί οι με την στήριξη άλλων γενναίων ηγετών στην Αθήνα και την Άγκυρα, του Πρωθυπουργού Παπανδρέου και του Πρωθυπουργού Ερντογάν, μπορούν να επιτύχουν μια λύση στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Βεβαίως, περιμένουμε όλοι μας οι φίλοι και σύμμαχοι να βοηθήσουν και αυτοί τους Προέδρους Ταλάτ και Χριστόφια. Πρέπει να υπάρχει νομίζω ενθάρρυνση και κίνητρο. Πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε για να έχουμε λύση την Κύπρο των συντομότερων Όσον αφορά τώρα την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η Τουρκία συνεισφέρει πάρα πολύ στις αποστολές αυτές στα Βαλκάνια, στην Αφρική και αλλού. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ που συζητάτε πάρα πολύ συχνά και ασκείται άδικη κριτική στην Τουρκία και στο πλαίσιο της έκθεσης για Τουρκία. Η έκθεση, η θέση με σχόλια της Τουρκίας είναι σαφής και επικοδομητική όσον αφορά την ΕΠΑ είναι άδικο να παρουσιάζεται η Τουρκία υπό οποιοδήποτε άλλο φως δεδομένη της δέσμευσης της και των πολλών συνεισφορών που έχει στην διατήρηση διεθνούς και περιφερειακής ε, σταθερότητας. Θα ήθελα να πω πως υπάρχει μια ισορροπία συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αμοιβαία διαφάνεια και συνεργασία. Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την ΕΠΑ καθώς και ε, την εμπλοκή μελών που δεν είναι μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ακολουθήσουν την διεύρυνση αυτής της στρατηγικής που ποτέ δεν ήταν προορισμένες να περιοριστούν στο Βερολίνο συν όπως σήμερα λανθασμένα πιστεύουμε. Υπάρχει λοιπόν ένας βαθμός περαιτέρω διαφάνειας που θα πρέπει να υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ΝΑΤΟ και όχι αυτή η στενή ερμηνεία και αντιμετώπιση του ΝΑΤΟ. Η ίδια περιοριστική φιλοσοφία ισχύει όσον αφορά την εμπλοκή συμμάχων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι σύμμαχος εντός του ΝΑΤΟ που είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στις επιχειρήσεις ΕΠΑ. Παρόλες τις ελλείψεις η Τουρκία είναι η χώρα η οποία συνεισφέρει περισσότερο στις επιχειρήσεις ΕΠΑ που δεν είναι μέλος της Ένωσης. Οπότε υπάρχει στήριξη από μια χώρα υποψήφια και σύμμαχο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την γενικότερη στρατηγική συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το να λέμε ότι την μπλοκάρει αυτή τη συνεργασία η Τουρκία δεν ανταποκρίνεται στα γεγονότα και τις εξελίξεις. Αναμένουμε λοιπόν οι λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για αυτή τη συνεργασία να γίνουν σεβαστές. Βεβαίως η Τουρκία, επειδή είναι πολύ σημαντική χώρα σε δύσκολη γεωγραφική περιοχή, αντιλαμβάνεται πως η γεωγραφία της ε, σημαίνει πως έχει κάποιες επιπλέον ευθύνες. Σε αυτό τον γεωγραφικό χώρο η Τουρκία παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον διαπολιτισμικό διάλογο. Είμαστε άλλωστε το ανατολικότερο κομμάτι της Δύσης και το δυτικότερο κομμάτι της Ανατολής. Και ως μια κοσμική ευρωπαϊκή δημοκρατία με κατά βάση μουσουλμανικό πληθυσμό παίζουμε το ρόλο του παραδείγματος, αν θέλετε, σε πολλές άλλες γειτονικές χώρες. προβάλλουμε τις ε, καθολικές μας αξίες και αποτελούμε εμπόδιο στην πόλωση. 1,5 δισεκατομμύριο μουσουλμάνοι ανά τον κόσμο παρακολουθούν από κοντά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Όταν λάβαμε ημερομηνία έναρξης ε, των συνομιλιών 17 Δεκεμβρίου 2004, εδώ στις Βρυξέλλες, στην Σύνοδο, υπήρχαν 430 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Οι 300 από αυτούς ήταν από μουσουλμανικές χώρες. Οπότε η διαδικασία αυτή παρακολουθείται στενά. Και η Τουρκία αντιλαμβάνεται πως έχει να παίξει ένα ρόλο. Ένα ρόλο που θα δημιουργήσει καλύτερο διάλογο και πολιτισμικές ανταλλαγές. Ο αριθμός ε, των μουσουλμάνων που ζουν στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει φτάσει σχεδόν τα 25 εκατομμύρια και αντιλαμβανόμαστε πως το μήνυμα που πρέπει να στείλετε στους μουσουλμάνους πολίτες σας, ανθρώπους που γεννιούνται εδώ, σε διάφορα κράτη-μέλη που είναι ψηφοφόροι σας, καταναλωτές σας, φορολογούμενοι, πρέπει να λάβουν λοιπόν το σωστό μήνυμα. Το να ξαναπροσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε το τείχος του Βερολίνου στους δρόμους της Ευρώπης και να χωρίσουμε τώρα το εσωτερικό των κρατών μελών δεν θα βοηθήσει κανέναν. Η οικονομία της Τουρκίας είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας. Αυτή τη στιγμή είναι η έκτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, 15η μεγαλύτερη στον κόσμο. Ως μέλος των G20 διαμορφώνουμε την παγκόσμια οικονομία με την τέταρτη μεγαλύτερη εργατική δύναμη στην Ευρώπη με μέση ηλικία τα 28. 65% των Τούρκων είναι κάτω από τα 35 έτη. Σημαντικό, αυτό σημαντική συνεισφορά που ε, έχει να κάνει η Τουρκία μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά τα ενεργειακά, η Τουρκία είναι διεθνής κόμβος για 70% των πόρων που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι είτε, είτε ανατολικά με συγχωρείτε, είτε νότια της ε, Τουρκίας ή και στα βόρεια. Επίσης, με τη Συμφωνία Ναμπούκο αποτελέσαμε μέρος της ενεργειακής λύσης και παραμερίσαμε μία από τις σημαντικότερες ε, δυσκολίες και κρίσεις όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. στηρίζουμε και άλλα έργα, όπως τη διασύνδεση Ελλάδας, Τουρκίας, Ιταλίας για φυσικό αέριο. Επίσης χτίζουμε αγωγούς για να περάσει αργό πετρέλαιο από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο. Γι' αυτό η Τουρκία θα συνεχίσει να παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, Μπορώ να σας πω πω ανακοινώσαν πρόσφατα από κοινού με την Κομισιόν πως θα ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει για τι συμφωνίε επανεισδοχή, αρκεί η συμφωνία να βασίζεται στο μοίρασμα του βάρου. Αντιλαμβανόμαστε πως είναι κοινό πρόβλημα αυτό και πρέπει να βρεθεί μια λύση από κοινού. Βεβαίω πρέπει να μα ενθαρρύνει και να μα στηρίξει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, γιατί όταν κάνει συμφωνίες με τρίτες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλαμε και εμείς να εμπλεκόμαστε και να έχουμε τις ίδιες συμφωνίες με χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Γεωργία και τα λοιπά. Αλλά τουλάχιστον τώρα έχουμε μια καλύτερη αντίληψη. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε κρατήσει γύρω στους 800.000 ανθρώπους σε τουρκικό έδαφος από αυτές τις χώρες. Πέρσι μόνο κρατήσαμε 65.000 άτομα και αντιλαμβανόμαστε πως με την ενισχυμένη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ο αριθμός αυτός θα διπλασιάζονταν ή τριπλασιάζονταν. Οπότε αναμένουμε την συνέχεια των συνομιλιών με τον Επίτροπο Μπαρόχτε. Ήμουν στη Στοκχόλμη, συναντήθηκα και με τον, ε, την μέλουσα Επίτροπο Σεσίλια Μάλμστρομ και ελπίζουμε το κοινό αυτό πρόβλημα να μην ε, αφαιθεί μόνο στην Ελλάδα και την Τουρκία και οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσουν στο να προλάβουμε τη λαθρομετανάστευση και να διασφαλίσουμε πω οι άνθρωποι που με κάποιο τρόπο έφτασαν μέχρι την Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη να ξαναστέλνονται σπίτι τους με ανθρώπινο τρόπο. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ο ισχυρότερο σύμμαχό σα στην καταπολέμηση διεθνού τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία είναι ένα ζήτημα που το γνωρίζουμε καλά. Ήμασταν θύματα της τρομοκρατίας του ΠΚΚ τι τελευταίε τρει δεκαετίε και είχαμε 40.000 νεκρούς. Το ΠΚΚ για μας είναι ότι η Αλκάιντα για τις υπόλοιπες δυτικές χώρες και αντιλαμβανόμαστε πως για να τελειώσει αυτό το κοινό πρόβλημα πρέπει να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε και τα πολιτισμικά δικαιώματα όμως των διαφόρων εθνοτήτων. Γι' αυτό είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος μιας κυβέρνησης στην Τουρκία που ξεκίνησε αυτή τη δημοκρατική πρωτοβουλία. Αντιλαμβανόμαστε πως κάποιες ομάδες στην Τουρκία είχαν δυσκολίες όσον αφορά τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Και δεν ήταν μόνο μία ομάδα. Πολλές διαφορετικές ομάδες. Δεν ήταν μόνο οι Κούρδοι, όχι μόνο οι Αρμένοι, όχι μόνο οι Έλληνες Ορθόδοξοι, όχι μόνο οι Σύριοι, όχι μόνο οι γυναίκες, όχι μόνο οι εργαζόμενοι, πολλές ομάδες. Είχαν προβλήματα με τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Δεν είμαι υπερήφανο για το ότι εκτελέστηκαν πριν από, πριν από 50 χρόνια πρωθυπουργοί στη χώρα μου μετά από πραξικοπήματα. Πριν από 30 χρόνια καίγαν τα βιβλία του Κάφκα, γιατί λέγαν πως ήταν κομμουνιστικά. Α, μην ξεχνάτε, ο πρωθυπουργό μου συνελήφθη πριν από 10 χρόνια για μία ανάγνωση ενός ποίηματος και ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό έχουμε ιδενική ανοχή στα βασανιστήρια σε τέτοιες συμπεριφορές και Θέλουμε να δούμε μια αύξηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του κάθε ενός πολίτη χωρίς καμία διάκριση με βάση εθνικότητα, θρησκεία, ιδεολογία, οτιδήποτε. Πιστεύουμε πως όλοι οι πολίτες της Τουρκίας πρέπει να ζουν με δημοκρατικά δικαιώματα και είναι η υπόσχεσή μας προς το έθνος μας να αυξήσουμε τις δημοκρατικές ελευθερίες. Αλλά για να επιτύχει αυτό στην, για να επιτύχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία, χρειαζόμαστε την δική σας στήριξη στην καταπολέμηση της θερμοκρατίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συνένεση στην χώρα μας για να αυξηθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα. Βεβαίως, η Τουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί εταίρο σας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων. Και όσον αφορά την αποφασιστικότητά μας για να συνεχίσουμε τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις, φέτος ξεκινάμε αποφασιστικά. Ξεκινήσαμε με ένα εθνικό πρόγραμμα την 1η Ιανουαρίου που αναφέρει το τι σκοπεύουμε να κάνουμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ένα έγγραφο 300 σελίδων υπάρχει και στο ίντερνετ στα αγγλικά. Στις 8 Ιανουαρίου για πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια, από όταν δηλαδή ζήτησε να ενταχθεί στην ΕΟΚ η Τουρκία, έχουμε έναν υπουργό που ασχολείται μόνο με τα ευρωπαϊκά και είναι επικεφαλής διαπραγματευτής. 16 Ιανουαρίου, μετά από τέσσερα χρόνια, ήρθε ο Τούρκος Πρωθυπουργό της Βρυξέλλης να συναντήσει τον κύριο Μπαρόσο. Τον Φεβρουάριο είχαμε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και τον Μάρτιο ήρθε εδώ πέρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Σε μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι πριν από 10 χρόνια φοβούνται να παραδεχτούν πως είναι Κούρδοι έχουμε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές ε, στην κρατική τηλεόραση στα κουρδικά 24 ώρες την ημέρα. Έχουμε επίσης μια επιτροπή ισότητας στο κοινοβούλιο μας. Δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ για το έργο της Νοτιοανατολικής Μικρασίας. Περάσαμε την νομοθεσία που πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για τις διαπραγματεύσεις. Αλλάξαμε το δασμολογικό μας δίκαιο, μειώσαμε τους ε, φόρους μας. Ε, επίσης θα δικάζονται οι στρατιωτικοί στα πολιτικά δικαστήρια. Έχουμε μια στρατηγική εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων στην δικαιοσύνη που έτυχε εκτίμηση από την Κομισιόν και θα ανακοινώσουμε νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Κάναμε πολλές αλλαγές για το περιβάλλον για να ξεκινήσει το κεφάλαιο του περιβάλλοντος 31 Δεκεμβρίου επί Σουηδικής Προεδρίας. Αλλάξαμε το φορολογικό κώδικα για να ξεκινήσει το κεφάλαιο της ε, φορολογίας στις τελευταίες ώρες της Τσεχικής Προεδρίας. πρωτομαγιά ορίστηκε αργία για τους ε, εργάτες. Ο Ναζίμ Χικμέτ επανέκτησε την υπηκότητά του, την οποία είχε χάσει πριν από 40 χρόνια λόγω της κομμουνιστικής του ιδεολογίας. Δεν ισχυρίζομαι πως λύσαμε όλα μας τα προβλήματα και έχουν επιτύχει όλες οι μεταρρυθμίσεις, αλλά είμαστε σωστό δρόμο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Στην Τουρκία γινόμαστε πιο δημοκρατική, πιο διαφανής χώρα και πηγαίνουμε στο δρόμο στο να έχουμε τις ίδιες προδιαγραφές με τις δικές σας χώρες. Και νομίζω αυτό είναι αμοιβαία επωφελές. Καθώς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε αυτές τι μεταρρυθμίσει, διασφαλίζουμε πως οι χώρες μας γίνονται πιο δημοκρατικές, με μεγαλύτερη ευημερία, πιο σύγχρονες, αλλά διασφαλίζουμε πως αντιμετωπίζετε κι εσεί έναν συνομιλητή πιο αξιόπιστο, πιο ισχυρό σύμμαχο σε πολύ σημαντική περιοχή. Steps to fulfill as a part of the democratic initiative. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Όπως είπα έχουμε σημαντικές ε, πρωτοβουλίες. Ε, σκοπεύουμε να κάνουμε σχολές κουρδικών στα πανεπιστήμια. Νόμος θα υπάρξει για την καταπολέμηση των διακρίσεων, ανεξάρτητη αρχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία να αλλάζει το όνομα πόλεων όταν το ζητάει ο πληθυσμό. Επίση, μπορεί να χρησιμοποιείται στι προεκλογικέ εκστρατείε και γλώσσα άλλη πλην τη τουρκική, αρκεί βεβαίω να γίνεται σεβαστό το Σύνταγμα και ο πλουραλισμό. Αντιλαμβανόμαστε πω για αυτό το Σύνταγμα θα έχουμε πρόβλημα βεβαίω να ενταχθούμε στην Ένωση. Και ελπίζουμε να υπάρξει συνένεση και στο δικό μας κοινοβούλιο με την αντιπολίτευση για να καταλήξουμε σε ένα σύνταγμα πιο διαφανές. Ποιο είναι λοιπόν, ποια είναι η θέληση του λαού της ε, Τουρκίας. Ο λαός της Τουρκίας απολαμβάνει τον εκδημοκρατισμό της χώρας μας και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, μέχρι το 2017 η Τουρκία θα είναι η τρίτη πιο γρήγορα αυξανόμενη οικονομία του κόσμου μετά την Κίνα και την Ινδία και τα τελευταία 7 χρόνια τριπλασιάστηκε το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Ήταν γύρω στα 3.000 δολάρια το 2000 και τώρα έχει φτάσει σχεδόν τα 11.000 δολάρια. Επίσης φτάσαν τα τελευταία 85.000 χιλιόμετρα τα τελευταία 85 χρόνια είχαν στη 6.000 χιλιόμετρα δρόμου. Εμείς, η κυβέρνησή μα, φτιάξαμε 9.000 χιλιόμετρα δρόμων ένα τέταρτο όλων των σχολείων, ένα τέταρτο όλων των νοσοκομιακών κλινών έγιναν επί κυβερνησής μας. Οπότε η Τουρκία γίνεται μια καλύτερη χώρα για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας και για να στείλετε και εσείς τα παιδιά σας για τουρισμό. Οπότε, η συνέχεια των συνομιλιών ένταξης είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ που με ακούσετε. Είμαι σίγουρος πως υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και θέλω να αφήσω και λίγο χρόνο για να δεχτώ ερωτήσεις. Και θα ήθελα να μάθω κι εγώ από εσά και να μεταφέρω μηνύματα στην πατρίδα μου. Ευχαριστώ. Caro Ministro, Υπουργέ, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την παρέμβασή σας, ε, που ήταν ε, πολύ πλούσια παρέμβαση ε, και πολύ σαφής. Πρέπει να το πω και αυτό. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα έχουν να θέσουν πολλές ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως να θέσω κάποιους κανόνες πάρα αυτά. Η συζήτηση θα ξεκινήσει με τη Ρία Όμεν Ρούιτε, την εισηγήτρια, και βλέπω ότι έχω 18 αιτήσει για παρεμβάσεις. Ο Υπουργός Φυσικά δεν έχει απεριόριστο χρόνο. Στις 4.30 ώρα θα πρέπει να φύγει. Ίσως ε, θα μπορούσε να μείνει ένα-δύο λεφτά παραπάνω. 4.30 γενικά θα πρέπει να φύγει. Σας καλώ όλους να είσαστε λακωνικοί, ούτω ώστε όλοι να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Όλοι όσοι το ζήτησαν. Δύο λεπτά λοιπόν έχει ο καθένας σας για να παρέμβει. Θα ξεκινήσει η συγγήτρια, η κυρία Όμεν Ρούιτεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω πως σέβομαι τον ανοιχτό και έξυπνο τρόπο με τον οποίο ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στις ανησυχίες που έχουμε οπωσδήποτε. Και θα ξεκινήσω με την ε, εξωτερική πολιτική. Ε, τα συζητήσαμε και το πρωί, τα είπαμε και με τον ε, κύριο Μπροκ ε, σήμερα το πρωί και σε σχέση με τη συνεργασία ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, όμως τώρα θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο άλλα σημεία που σχετίζονται άμεσα με την Τουρκία και τη σχέση με τους γείτονες. Πρώτα απ' όλα Αρμενία. Ευθύ εξ αρχής είχα πει πως το σημαντικότερο είναι για να ξεπεράσουν το παρελθόν η Αρμενία και η Τουρκία να ανοίξουν τα σύνορα. Τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν τώρα. Τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε ως εκπρόσωπος ε, της κυβέρνησης και της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ε, ομάδας του Κοινοβούλιο για να υπογραφούν αυτά τα πρωτόκολλα. Δεύτερον, σχέσεις με την Κύπρο. Ξέρω πως ε, χτες ε, είχαμε επίσκεψη του κυρίου Ταλάτη στη χώρα σας, μιλήσατε για τις συνομιλίες που υπάρχουν στο νησί για την επανένωση. Εσείς ο ίδιος είστε θετικός, αλλά ξέρουμε πως μπορεί να είστε θετικός, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Και δεν μιλάω τώρα για το πρωτόκολλο της Άγκυρας, υπάρχει αυτό στην έκθεσή μου, αλλά να φροντίσετε οι δύο κοινότητες να δώσουν, να κάνουν θετικά μηνύματα, το είπαμε αυτό και πέρσι, όπως και φέτος, για να έχουμε μια οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Κατόπιν, τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Θαυμάζω πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα στην χώρα σας, το πώς αντιμετωπίζετε τους Κούρδους, το πώς ανακοινώνετε ότι θα κάνετε κάτι. Ευαίσθητη υπόθεση, αλλά το κάνετε. Τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε για τους Αλεβίτες. Αλλά σας παρακαλώ να το κάνετε αυτό και για τους μη μουσουλμάνους. Γιατί εκεί πέρα έχετε κάνει θετικά βήματα στα λόγια, αλλά πρέπει να μεταφραστούν και σε νομοθεσία και να περάσουν από το Κοινοβούλιο. Και εκεί πέρα σας ζητώ να κάνετε κάτι. Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάμε για δικαιώματα γυναικών, γυναικών καταπολέμησης διακρίσεων κτλ. Μιλάω για τις εκστρατείε που κάνει η κυρία Γκιούλη, η κυρία Ερντογάν και πολλές άλλες γυναίκες για να προσπαθήσουν να αλλάξουν την οτροπία της κοινωνίας σας. Θετικό. Και η νομοθεσία είναι θετική, αλλά τι θα γίνει με την εφαρμογή στην πραγματικότητα έχετε σχέδια συγκεκριμένα. Πρέπει να επικεντρωθείτε έτσι ώστε αυτό το οποίο έχει γίνει νόμος να εφαρμοστεί και όλα στην πραγματικότητα. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, δεν θα μιλήσω όλα. Δεύτερη παρέμβαση θα είναι από την κυρία Φλότχ. Δύο μινούτι. Με... Έχετε δύο λεπτά, κυρία Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Μπαγκής για την προθυμία που έδειξε και το ότι είναι διαθέσιμος και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και στην Μικτή Επιτροπή. Νομίζω ότι έχετε, έχετε πολλούς λόγους να είστε υπερήφανος για την δημοκρατική σας προσήλωση που φαίνεται στις ε, σημαντικές μεταρρυθμίσεις που είναι ουσιώδεις για τη δημοκρατική αλλαγή και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει λοιπόν ε, εμείς οι Ευρωπαίοι ε, να μην σας υποστηρίξουμε, αλλά και εσείς οι Τούρκοι να μην δείξετε την απαραίτητη τόλμη. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Έχω τρεις Ερωτήσει ε, που συνδέονται άμεσα με τι διαπραγματεύσει και το άνοιγμα των κεφαλαίων. Το θέμα τη συνδικαλιστική ελευθερία που μπλοκάρει, γιατί το νομοσχέδιο για τα συνδικάτα μπλοκάρει το άνοιγμα του κεφαλαίου για την επασχόληση και τα κοινωνικά θέματα. Φαίνεται δύσκολη η ανέβρεση συνένεση. Πώ θα ε, αυτό το αδιέξοδο για σημαντικά θέματα συνδικαλιστικής ελευθερίας, δικαιώματος απεργία κτλ. Δεύτερον, συμφωνία επανειστοχής. Το Συμβούλιο και ε, ο Ήπατος ε, αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, έχουν υπογραμμίσει καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των ετών άσυλων στα σύνορα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων να συμπεριληφθούν στις συζητήσεις για τις συμφωνίες επανεισοχής. Επίσης, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ο Πρωθυπουργό εξήγηλε πριν από λίγους μήνες στο άνοιγμα αυτής της θεολογικής σχολής, κάτι που δεν έγινε, που κόλλησε τα πράγματα, γιατί έχουν αποτελματωθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπροκ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω διάφορες παρατηρήσεις εδώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ και τώρα, παρότι έχουμε ένα καινούριο κοινοβούλιο. Παρότι είμαστε καινούριο κοινοβούλιο, έχουμε μια πειραμένη συγγήτρια. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε παρότι δεν είναι παρόν κάποιος Σουηδό από του εκπρόσωπου τη Σουηδική Προεδρίας εδώ. Θα ήθελα να πω κάτι για την πολιτική ασφαλεία. Ο κ. Μπαγκή μίλησε για το ρόλο τη Τουρκία στην περιφέρειά του, στην γεωγραφική του ζώνη. Το θέμα που μας ενδιαφέρει εδώ όλους είναι πώς το θέμα του Ιράν θα εξελιχθεί. Σκέφτομαι την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κυρίου Ερντογκάν στο Ιράν. Έχω υπόψη μου επίσης την Τουρκία, η οποία βοηθάει για την εξαγωγή πυρηνικού υλικού. Δεύτερο σημείο. Όλα συνδέονται βέβαιως. Και όλα συνδέονται τελικά με το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Ίσως κάποια χειρονομία θα μπορούσε να γίνει στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας. Θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε κάποια πράγματα τη στιγμή που η χώρα σας θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ δεν ε, πηγαίνει όσο καλά θα έπρεπε, μας κοστίζει πάρα πολλά λεφτά και μας εμποδίζει, μας παρεμποδίζει από το να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε. Έχετε κάποιες ιδέες για αυτό το θέμα, για αυτές τις σχέσεις. Ίσως η Τουρκία θα μπορούσε να αποποιηθεί του δεύτερου ρόλου της στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ, ο κύριος Όουι. Χάουιτ. Ε, έχετε μεγάλη, πολύ μεγάλη φήμη από τη στιγμή που αναλάβατε το αξίωμα του βασικού διαπραγματευτή. Ε, νομίζω ότι υπάρχει πρόοδος μεταξύ μας, υπάρχουν θετικά μηνύματα. Ερωτήσεις, ε, καταρχάς. Από αυτό το 400 σέλιδο σε κείμενο, ε, εγώ πιστεύω ότι όντως θα πρέπει να κοιτάξουμε προς τα εμπρός, όχι και προς τα πίσω όπως η Κομισιόν. Ε, τους επόμενους 12 μήνες του 2010, τι πρόοδος περιμένετε να σημειωθεί για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Ε, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη μια διακομματική συμφωνία. Ε, εσείς και το κόμμα σας ε, ε, συχνά κατηγορείται την αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση α, κατηγορεί εσά. Είναι δύσκολο να περάσουν αυτέ τι μεταρρυθμίσει συνταγματικέ. Πώ θα μπορούσε να κινηθεί αυτό το θέμα στο εσωτερικό τη Τουρκία και να προωθηθεί. Ε, για την ελευθερία τη έκφραση. Ε, πιστεύω πραγματικά ότι οι περαιτέρω νομικέ αλλαγέ, παρότι είναι απαραίτητε, δεν είναι επαρκεί. Ποια είναι η άποψή σα για τις κατευθυντήριες γραμμές προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για κάποια τέτοια θέματα. Και ποια είναι η απόψή σας για τους ε, υψηλόβαθμους δικαστές που εμπλέκονται σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, ε, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Επίσης, πολλοί μίλησαν για το κουρδικό και το αρμενικό θέμα. Είναι δύσκολα θέματα. Ε, ότι η κυβέρνησή σας δεν θα μπορούσε να τα είχε προωθήσει, αλλά τα κατάφερε. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσει τι σας ε, βοήθησε για να, να σημειώσετε αυτή τη σημαντική πρόοδο. Γιατί αν το καταλάβουμε, ε, μπορούμε να καταλάβουμε και πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και σε άλλους τομείς πέρα από αυτούς. Ευχαριστώ κύριο Λάμστορφ. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνικός γιατί ήδη με πρόλαβε ο Ρίτσαρτ Χόουιτ για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι κάτι που το ακούμε από το 2004. Περιμένουμε λοιπόν τη δική σας απάντηση για το τι πρόοδος αναμένεται σε αυτό το θέμα. Και πού θα γίνει, πού θα σημειωθεί η καμπή. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και τις ε, σχέσεις με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή. Η αποστολή UPOL στο Αφγανιστάν έχει πρόσβαση σε στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών. Ναι ή όχι. Απλή μονολεκτική απάντηση. Έχει πρόσβαση στα δεδομένα της ISAF. Καλή συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, αλλά επί τόπου τι γίνεται. Επίσης μιλούμε για, το, για την ασφάλεια του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλές οι πολιτικές και θεσμικές συζητήσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε εμπράκτο πώς, ε, μεταφέρεται, πώς μεταφράζεται η συνεργασία. Έχει UPOL ε, πρόσβαση στι μυστικές πληροφορίες της ISAF ή σε άλλα δεδομένα ασφάλειας. Είπατε ότι η τουρκική οικονομία είναι εύρωστη και πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα χάσμα αναπτυξιακό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Το κατακεφαλήν ΑΕΠΣΕΣ είναι το ίμιση της ενώσης πριν την, γύρω στην διεύρυνση του 2004, ενώ ο πληθυσμός σας είναι πολύ μεγαλύτερος. Οπότε η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει πολύ περισσότερες προσπάθειες για να γεφυρώσει αυτό το κοινωνικό-οικονομικό χάσμα. Ο κύριος Βανόρντεν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερο ε, που σας βλέπω εδώ και πολύ εκτιμούμε τη σημασία της Τουρκίας που είναι ε, θεμελιώδη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, έχει αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη, ζωτικό ρόλο στον ενεργειακό κλάδο και έχει κρίσιμη γεωστρατηγική θέση ως μουσουλμανική χώρα. Θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος και έχουμε επίγνωση των ανησυχιών των πολιτών μας για θέματα μετανάστευσης και όχι κατά υπό το πρίσμα της κυρίας Φλότρ. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση για το Κυπριακό, γιατί γνωρίζω ότι αφενός η Κύπρο ε, είναι κάτι ξεχωριστό από το θέμα της Ένταξη της Τουρκίας, αλλά το Κυπριακό είναι ένα κόλλημα στην ε, συντέλεση πρόοδου. Τι μπορεί να γίνει ε, για, από τρίτους για την επίλυση του Κυπριακού, γιατί όλο με την Τουρκία. Οι υπόλοιποι όμως τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν την ε, επίτευξη λύσης. Τώρα, από τουρκική άποψη. Υπάρχουν κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, εδραίωσης της εμπιστοσύνης που μπορείτε να λάβετε εσείς. Για παράδειγμα, ε, μείωση της στρατιωτικής παρουσίας στο βόρειο του νησιού. Έτσι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα θετικότερο κλίμα για τις εκκρεμείς διαπραγματεύσεις που ίσως καταλήξουν σε αίσια έκβαση. Για κάτι διαφορετικό τώρα. Αναφέρθηκε το Αφγανιστάν. Και ο συνάδελφος Γκραφ Λάμστορπ ε, έθεσε μια πολύ σημαντική ερώτηση γιατί η Γιούπολ δεν έχει σχέση με την ε, πρόσβαση στι μυστικέ υπηρεσίε. Κανονικά έπρεπε να εκπαιδεύουν αστυνομικού, κάτι που δεν κατάφερα το κάνω, απέτυχε εκεί η Γιούπολ. Για το Αφγανιστάν όμω, το θέμα της ενίσχυσης των στρατευμάτων είναι ένα ζήτημα. Η Τουρκία πρόκειται να στείλει και άλλα στρατεύματα για να ενισχύσει τις προσπάθειες της ISAF στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση της πρώτης ομάδας. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Χατζηγεωργίου, παρακαλώ. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ εσάς εδώ στη συνεδρία, κύριε Μπαγής, Να σας πω ότι εμείς στην Κύπρο έχουμε ιδιαίτερους λόγους να παρακολουθούμε τα όποια θετικά βήματα κάνει η Τουρκία, η χώρα σας, προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και στην προσπάθεια σας για ένταξη. Θέλω να σας πω πολύ ειλικρινά ότι και τα παρακολουθούμε και τα σημειώνουμε. Όμως αυτό δεν μας επιτρέπει καθόλου να αγνοούμε το πόσο δρόμο έχετε ακόμα μπροστά σας να διανύσετε σε πολλά άλλα ζητήματα. Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε. Πιστεύω ότι υποστηρίξατε την υπόθεσή σας με σχετική υπερβολή σε σημείο που κινδυνεύσατε να την υποσκάψετε. Και θέλω να πω ότι η Κύπρος και εγώ προσωπικά θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την αισιοδοξία σας για επίλυση. Υποστηρίζομαι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μόνον εφόσον η Τουρκία συμβάλλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της επίλυσης και νομίζω ότι η κουβέντα που λέτε συχνά πυκνά ότι οποιαδήποτε λύση βρουν οι Κύπροι ηγέτες, οι δύο ηγέτες στην Κύπρο θα την υποστηρίξετε, είναι ως να βγάζετε την ουρά σας έξω από ένα πρόβλημα που δεν μπορείτε να το κάνετε. Έχετε εκεί 40.000 στρατό. Θέλω να πω κάτι και για αυτό που είπε, που τώρα μόλις ο κύριος Βανόρτεν και να το συνδυάσω με μια δήλωση δική σας προχθεσινή στο TRT channel της Στοκόλμης όπου είπατε, θα το πω στα αγγλικά όπως το βλέπω γραμμένο Έχουμε αλλάξει όλες τις διεθνείς ισορροπίες στο νησί χωρίς να αποσύρουμε ούτε έναν στρατιώτη δίνοντας όμως ειρήνη στο έδαφος. χωρί και χωρίς να δώσουμε ούτε σπιθανή εδάφους, μάλλον, συγγνώμη. Αναφορικά με τις σχέσεις της με τις γυναικές χώρες, συνοψίζεται στις λέξεις μηδανικά προβλήματα και θέλουμε να το χειροκροτήσουμε. Πώς συνάδει όμως αυτό με την πολιτική της συντήρησης από πλευράς της Τουρκίας του στάτους κβό της κατοχής, δεν συνεισφέρεται ουσιαστικά στην επίλυση του Κυπριακού με απόσυρση του στρατού. Υιοθετώντα τη λογική τη επιλεκτική στάση έναντι των γειτονικών χωρών κλείνω με μια φράση, και των Ευρωπαίων εταίρων, όπω παραδείγματος χάρη με την φύ εφαρμογή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου, δεν είναι η ίδια η Τουρκία που δεν βοηθά την πρόοδο των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων. Αφήσουμε 10 λεφτά στον Υπουργό για να απαντήσει σε αυτόν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Συστήνω στους συναδέλφους να περιορίσουν ε, το χρόνο της παρέμβασής τους, γιατί αλλιώς κάποιος ε, δεν θα μιλήσει και αυτό θα ήταν πολύ δυσάρεστο για εκείνον. Well, I would like to thank... Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για τα επικοδομητικά του σχόλια, τις κριτικές και τις ερωτήσεις και απορίες τους. Σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα με την Αρμενία. Αν πριν από πέντε χρόνια μου έλεγε κάποιο ότι ο Πρωθυπουργό τη Τουρκία θα μπορούσε να υπογράψει πρωτόκολλο με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Αρμενία, δεν θα τον πίστευα. Και όμω τα καταφέραμε. Κάτι που δείχνει ότι η Τουρκία θέλει την ειρήνη. Και όταν είπαμε μηδενικά προβλήματα με του γείτονε, καμία χώρα πριν από 7 χρόνια δεν πίστευε ότι θα το καταφέρναμε. Σήμερα όμω ε, έχουμε αυξήσει κατά 300% το, ξένο μας, το διεθνές μας εμπόριο και έχουμε αυξήσει κατά 50% το διεθνές εμπόριο με τους γειτονές μας. Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να ενισχύσει την σχέση της με τους γειτονές της και η πολιτική αυτή έχει αποδώσει καρπούς. Αν πριν από 10 χρόνια μου έλεγε κάποιο ότι θα έρθει μια μέρα όπου ο Πρωθυπουργό της Ελλάδας θα γίνει μάρτυρα, θα είναι μάρτυρας ή κουμπάρος στο γάμο της κόρης του Τούρκου Πρωθυπουργού. Ούτε και αυτό θα το πίστευα. Θα έλεγα πίστευτο. Και όμως ακόμη και αυτό το είδαμε τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός Καραμάλη ήταν ο μάρτυρας στο γάμο της κόρης του Ερδογάν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει, έχουν αυξηθεί οι αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από 2 σε 11. Έχουμε προσπαθήσει να αποφύγουμε τη διπλή φορολόγηση και ε, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας που έχει βασικό μέτοχο την Εκκλησία της Ελλάδας είναι ιδιοκτήτρια τραπεζών τουρκικών και αξίας δισεκατομμύριων με χαρτοφυλάκιο δισεκατομμύριων. Έχουν αλλάξει λοιπόν όλα αυτά τα ήθη και έθιμα στις διεθνείς σχέσεις. Πριν από 10 χρόνια 300.000 ε, ε, στρατιώτες είχαμε αναπτύξει τα σύνορά μας με τη Συρία, γιατί η Συρία υποστήριζε την τρομοκρατία του ΠΚΚ. Σήμερα η ίδια αυτή χώρα, η Συρία, συνέλαβε τρομοκράτες του ΠΚΚ και τους εξέδωσε, τους παρέδωσε στο τουρκικό δικαστικό σύστημα. Και μάλιστα τώρα αποφασίσαμε να άρουμε τις κυρώσεις σε θεωρήσεις. Και μάλιστα από 200 εκατομμύρια έγινε 2 δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια το ο, ύψος του εμπορίου μας με την, Τουρκία, με την Συρία. Συγγνώμη. Και στη σχέση μας με την Αρμενία υπάρχει τεράστιο δυναμικό. Και ήταν πολύ εύστοχη η ερώτηση της Συρία. έχουμε την πρόθεση να οικοδομήσουμε καλύτερε σχέσει με όλε τι γειτονικέ μα χώρε συμπεριλαμβανομένε τη Αρμενίας. Αλλά θα πρέπει να θυμάστε γιατί είχε κλείσει η Τουρκία τα σύνορά της με την Αρμενία. Παρόλο που ήταν μια από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Αρμενίας μετά την κατάρρευση της Σοβιετική Ένωσης. Κλείσαμε τα σύνορα εξαιτίας της εισβολής στο Καραμπάχ. Έπρεπε να δείξουμε αλληλεγγύη προς τη γειτονική χώρα του Αζερμπαϊτζάν. Τώρα περιμένουμε από την ομάδα του Μίνσκ, κυρίως στη Ρωσία και τις Ηνωμένε Πολιτείε και τη Γαλλία, για να βρουν μία λύση και να ξεφύγουμε από το διέξοδο στις ε, συνομιλίες για το Καραμπάχ. Πιστεύω ότι το Παρίσι, η Γόσιγκτον και η Μόσχα, θα συνεργαστούν, αν συνεργαστούν καλά, θα καταφέρουν πολύ εύκολα μία συμφωνία για το Καραμπάχ. Κάτι που θα διευκολύνει και εμάς και θα μας επιτρέψει να κυρώσουμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση το πρωτόκολλο με την Αρμενία. Και θα δημιουργήσει και ένα καλύτερο κλίμα, πιο πρόσφορο, για να κυρώσει και η Αρμενική Βούλη το πρωτόκολλο. Γιατί και οι δύο χώρες είναι απρόθυμες, ε, διστακτικέ και περιμένουν πρόοδο. Αλλά θέλουμε ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Νικολά Σαρκοζή και ο Μετβέντεφ να επιδείξουν ε, πρωταγωνιστικό ρόλο και ε, να δώσουν κίνητρα στους, ε, στον Αλίεβα και τον Αλίεβα Σαρκισιάν για να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Ένα ζήτημα που έθεσαν πολλοί ευρωβουλευτές. Θα δώσω μια γενική απάντηση για το θέμα της Κύπρου. Κάποιο είπε για μια χειρονομία. Αλλά αυτό που κάνω από το 2002 είναι μια ολόκληρη σειρά χειρονομιών. Τον Ιανουάριο του 2003, όταν ο Πρωθυπουργό συνάντησε στον Ταβό στον Γενικό Γραμματέα Κόφη Ανάν και του ζήτησε να ξεκινήσει τον τέταρτο γύρο των διαπραγματεύσεων, η πρώτη απάντηση του Γενικού Γραμματέα Ανάν, και ήμουν παρόν εκεί, ήταν Κύριε Πρωθυπουργέ, τρει φορέ το έχω προσπαθήσει και τρει φορέ απέτυχα. Δεν θέλω να αποτύχω και τέταρτη φορά. Τότε ο Πρωθυπουργό Ερδογκάν έκανε μία υπόσχεση. Είπε: Σα υπόσχομαι, κύριε Γενική Γραμματεύ, ότι εμείς θα, θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε και τους Ελληνοκύπριους και τους ε, Τουρκοκύπριους και θα κάνουμε προσπάθειες για να επιτύχει ε, η συνομιλία σας. Και όταν χρειάστηκε να βάλουμε τις αδρές γραμμές αυτού του σχεδίου, η Τουρκία πρότεινε, έκανε προτάσεις για θέματα που ήταν πολύ δύσκολα για συμφωνία και μάλιστα αφήσαμε κάποια κενά για να τα συμπληρώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Και όταν στο Μπούργενστοκ καταρτίστηκε το σχέδιο, ήμουν και εγώ μέλος τότε της τουρκικής αντιπροσωπείας και εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να πετύχουμε μία λύση. Πιστέψτε με, το σχέδιο Ανάν ούτε και για μας ήταν τέλειο, αλλά τουλάχιστον ήταν δίκαιο και ισορροπημένο. Αλλά και, αυτό, και από αυτό χρειάστηκε να παραιτηθούμε. Αν είχε εγκριθεί το σχέδιο Ανάν, ο αριθμός των τουρκικών στρατευμάτων που θα έμεναν στο νησί αυτή τη στιγμή ήταν 650 στρατιώτες. Μόνο 650 θα έμεναν για μία πενταετία αν είχε εγκριθεί το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και μετά την πέμπτη χρονιά θα διοργανώνονταν δημοψήφισμα μετά από μία πενταετία θα διοργανώνονταν δημοψήφισμα και θα μειώνονταν και τα ελληνικά στρατεύματα σε 900 στρατιώτες. Αν λοιπόν όλες οι άλλες χώρες που έχουν στρατεύματα στο νησί, αν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι διατεθειμένε να αποσύρουν τα δικά τους στρατεύματα, ε, να το εξετάσουμε και αυτό, να εξετάσουμε αυτή την ιδέα. Σχόλια εκτός μικροφώνου δυστυχώ. Ναι, ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε Εντάξει, όταν μιλάμε για τα δικά σα στρατεύματα είναι εθνική κυριαρχία. Όταν μιλάμε για τα δικά μα στρατεύματα θέλετε χειρονομία. Εάν είναι να κάνουμε χειρονομία, κάνουμε χειρονομία όλε οι πλευρέ. Πάντω θα πρέπει να υποστηρίξουμε του δύο προέδρου, ε, Χριστόφια και Ταλάτ, προκειμένου να καταλήξουν σε αποδεκτή λύση. Γιατί με το σχέδιο Ανάν είχαμε δυσκολίε. Ο Πρωθυπουργό Ερντογκάν έκανε κάποιε προσφορέ στον ε, πρόεδρο Παπαδόπουλο και πρωθυπουργό Καραμαλή για αναβολή των συνομιλιών, αλλά είχε, κάνει υπόσχεση, είχε δώσει υπόσχεση προ τον ε, Γενικό Γραμματέα Ναν και υποστήριξε το σχέδιο Ναν. Τώρα για την εκστρατεία του σχεδίου. Ο Ερντογάν ήταν ο ηγέτης που δημόσια υποστήριξε το σχέδιο Ανάν. Παρά την αντίθεση του Ντεκτάς στην Τουρκία και την, ε, στην τουρκική πλευρά μάλλον, τουρκοκυπριακή και του Παπαδόπουλου στην ελληνοκυπριακή. Και το 65% των Τούρκων ψήφισαν ναι στο σχέδιο, ενώ οι Ελληνοκύπροι 76% είπαν όχι στο σχέδιο. Είπαν όχι στην ε, συνύπαρξη με τους ε, Τούρκους, είπαν όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν όχι στις εκκλήσεις ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Εμείς όμως δεν τα παρατήσαμε. Είπαμε εντάξει αυτό δεν πέρασε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Στις 26 Απριλίου 2004 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση. Και τότε, για να εφαρμόσουμε το πρωτόκολλο της Άγκυρας, ζητούσαμε, το μόνο που ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εφαρμόσει την ηλυμένη της απόφαση. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να θέσει τέρμα στην απομόνωση των Κυπρίων του Βορείου Τμήματος. Κανεί δεν αναγνωρίζει από εμά την Ταϊβάν, αλλά όλοι έχουμε εμπορικέ σχέσει με την Ταϊβάν. Γιατί δεν γίνεται το ίδιο και με του τουρκου για να τεθεί ένα τέρμα στην απομόνωσή του. Σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, από τι 27 χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο μία έχει άμεσο εμπόριο με το βόρειο τμήμα. Δεν θα πρέπει να μείνει μόνη τη αυτή η χώρα. Και αυτή η μόνη χώρα είναι η Νότια Κύπρος. Οι Ελληνοκύπροι έχουν ελεύθερο εμπόριο και ελεύθερη διακίνηση προς το βόρειο του Ματουνισιού, αλλά θέλουν οι υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια. Αυτό είναι άδικο. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις συνεχείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Σε ό,τι αφορά το, σχέ, το νομοσχέδιο για το συνδικαλιστικό κίνημα και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Θέλουμε να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες μας με εμπορικούς και επιχειρηματικούς και συνδικαλιστικούς κύκλους. Χθε ήμουν σε συνομιλίες και με τις δύο πλευρές και για να ξεκινήσει να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε ένα συνδικαλιστικό νόμο που θα τηρεί τις προδιαγραφές του κοινοτικού δικαίου. Αλλά πρώτα φυσικά θα πρέπει να καθίσουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων οι ηγέτες ε, αρχηγοί του επιχειρηματικού κύκλου και του συνδικαλιστικού κινήματος και αυτό θα γίνει στο νέο γύρο διαπραγματεύσεων που ευελπιστούμε ότι θα γίνει σύντομα προκειμένου να ανοίξει και το σχετικό κεφάλαιο. Για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Η Χάλκη δεν έκλεισε με απόφαση της κυβέρνησής μου. Η Χάλκη έκλεισε εξαιτία ε, δικαστικής απόφασης. Και τώρα εξετάζουμε το νομικό καθεστώς. Πώς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν θα πρέπει να τροποποιήσουμε το νόμο, το σύνταγμά μας ή ένα απλό κανονισμό. Είναι μια τεχνική διαδικασία, αλλά επεξεργαζόμαστε αυτές τις λύσεις. Και επίση δεν υπάρχει μόνο θέμα ασφάλεια. υπάρχει θέμα και χριστιανικών κοινοτήτων, μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Γιατί κάποιο μίλησε για τις μειονότητες στην Τουρκία. Προσπαθούμε να επιλύσουμε και τα δικά του προβλήματα. Χθε στη Στοχόλμη συναντήθηκα με ηγέτε της ασυριανής Έχουν και αυτοί θέματα και τα συζητούμε. Σε ό,τι αφορά το ρόλο μα με το Ιράν. Νομίζω τα παλιότερα σύνορα του κόσμου είναι αυτά της Τουρκίας και του Ιράν που από το 1639 δεν έχουν αλλάξει ούτε ένα εκατοστό. Και πρέπει να έχουμε επαφές με το Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να, για να αποτρέψουμε άλλο πόλεμο στην περιοχή και θα συνεχίσουμε στην προσπάθεια ανέβρεσης λύσης. Πιστέψτε με, αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα, οι πρώτοι που θα ανησυχούσαμε θα ήμασταν εμείς. Αλλά Μιλούμε με τους Ιρανούς φίλους και γείτονες και για να μιλήσει κανείς με τέτοιου Ιρανούς φίλους και γείτονες θα πρέπει να έχει διαφορετικά επικοινωνιακά προσόντα από αυτά που χρησιμοποιείται εσείς στην Κεντρική Ευρώπη. Ίσως η ανατολικό-ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι πιο δόκιμη, λογική όταν επικοινωνεί κανείς με το Ιράν. Φυσικά θέλουμε λύση και στο πρόβλημα αυτό. για το θέμα της συμμετοχής δικαστών σε κοινοτικά προγράμματα. Έχουμε πολλά προγράμματα κατάρτισης δικαστών και μάλιστα το δικαστικό σώμα είχε πολύμινες συζητήσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να καταλήξουμε σε μια περιεκτική και συνενετική λύση για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου. Και τώρα προετοιμάζουμε το σχέδιο δράσης αυτού του εγγράφου στρατηγικής που θα αλλάξει τελείως το δικαστικό τοπίο και την απονομή δικαιοσύνη στην Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, είμαι αισιόδοξο. Το 2010 είναι η μόνη χρονιά στην Τουρκία που δεν θα έχουμε εκλογέ. Ευκαιρία λοιπόν να θεσπίσουμε και να εφαρμόσουμε κάποιε μεταρρυθμίσει. Εσεί οι πολιτικοί γνωρίζετε ότι δύσκολο είναι να περάσουν οδυνηρέ μεταρρυθμίσει σε χρονιέ που γίνονται εκλογέ. Μια και το 2010 δεν θα έχουμε εκλογέ, Ευελπιστούμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεργαστούν μαζί μας όπως έγινε το 2002 και το 2005 και θα υλοποιήσουμε από κοινού αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της ΕΠΑ, το μόνο που θέλει η Τουρκία είναι ίση μεταχείριση, δίκαιη μεταχείριση. Είμαστε για πάνω από 50 χρόνια μέλος του ΝΑΤΟ και έχουμε το δεύτερο σημαντικότερο στρατιωτικό σώμα στο ΝΑΤΟ. Θέλουμε τα ίδια προνόμια με τους υπόλοιπους συμμάχους του ΝΑΤΟ στα πλαίσια της ΕΠΑ. Θέλουμε και εμείς να γίνουμε τμήμα της ασφάλειάς σας. Δεν θέλουμε να είμαστε τμήμα του προβλήματος, αλλά τμήμα της λύσης από κάθε άποψη. Για τις ε, κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Εγώ ανέφερα ότι το κατακεφαλήν εισόδημα ε, στην Τουρκία από 3.000 ε, δολάρια έφτασε στα 11.000 δολάρια μέσα σε 7 χρόνια. Αν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα είχατε μια τόσο έντονη οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, πέστε μου το. Ε, δουλεύουμε για να κλείσουμε το κενό και τη διαφορά που μας χωρίζει από εσά. Και το γεγονός ότι ο λόγος αυτός μειώνεται. Ε, το γεγονός ότι οι άμεσες οι επενδύσεις που ερχόταν στην Τουρκία πριν από το 2003 ήταν περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, ενώ τώρα είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αυτή η κοσαπλάσια αύξηση είναι ένα σαφέστατο δείγμα ότι κλείνει αυτό το χάσμα της ψαλίδας στο κοινωνικό-οικονομικό τομέα και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Για τα περισσότερα στρατεύματα στο Αφγανιστάν ε, θα υπάρξει αύξηση των στρατευμάτων αλλά μετά την πρόσφατη αναγγελία του Πρόεδρου Ομπάμα αν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ αποφασίσουν να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο Αφγανιστάν και στα προγράμματα αυτά, η Τουρκία φυσικά θα υποκληθεί στην γνώμη της πλειοψηφία. Είμαστε όλοι στο ίδιο κλαμπ και όλοι θα πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες ε, που μας συνενώνουν. Όπως δημοκρατία, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία λόγου, γι' αυτό όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν είναι μια πολύ σημαντική χώρα για μας. Πήγα μαζί με τον Πρωθυπουργό μου στο Αφγανιστάν και με εξέπληξε η φτώχεια και οι δυσκολίες τις οποίες είδα τα ίδια μου τα μάτια. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε το Αφγανιστάν ε, και να, το βοηθήσουμε για να επιλύσει τα προβλήματά του. Νομίζω ότι αρκούν αυτά, μπορώ να σταματήσω. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Σαλαφράγκα. Θα σας κλέψουμε, κύριε Υπουργέ, λίγο χρόνο. Θα σας αναγκάσουμε να καθίσετε λίγο περισσότερο μαζί μας για να δώσετε απαντήσεις στους συναδέλφους. Κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Υπουργό που ήρθε και αφιέρωσε τον χρόνο του στην Επιτροπή μας για να μας εξιστορήσει τις ε, εξελίξεις και την εντυπωσιακή πρόοδο που πραγματοποιεί η χώρα του, όπως ε, μας είπε και στην έκθεσή της η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Θα κάνω μια ερώτηση κάπως προκλητική. Η πρόοδος αυτή αναφέρθηκε σε κάποιες τροποποίησεις σε συνταγματικά θέματα, ποινικά, ελευθερία των γυναικών, ελευθερία πληροφόρησης και ούτω καθεξής. Μας δίνεται την εντύπωση από κάποιες δηλώσεις ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα αυτό προεδρεύεται του Συμβουλίου, που έκανε σήμερα έναν απολογισμό ή είπατε εκπρόσωπο σήμερα μας είπε ότι το 2009 μόνο ένα, ένα κεφάλαιο έκλεισε από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Έχω την αίσθηση ότι ε, όταν ξεπερνάμε ένα εμπόδιο με την Τουρκία βγαίνει άλλο εμπόδιο. Θυμά, μου θυμίζει το μύθο του Σισίφου που είχε καταδικαστεί από τους θεούς να ανεβάζει ένα βράχο στο, στην κορυφή του βουνού και μετά τον άφηνε να πέσει στους, στις παρυφές και αυτό και από την αρχή. Αυτό μου θυμίζει η τακτική της Τουρκίας. Αυτή όμως η συμπεριφορά των εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μήπως ε, υπονομεύει την αποφασιστικότητα της τουρκικής κυβέρνησης για συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Και τι γίνεται με τους Τούρκους πολίτες. Τι επίχυση έχει αυτή η κατάσταση στον τουρκικό λαό. Μήπως υπάρχει κάποια κόποση από τις ε, διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η υποστήριξη της ενταξιακής διαδικασίας ε, στην ε, Ένωση έχει μειωθεί σημαντικά. Ποια είναι η σημερινή θέση των Τούρκων πολιτών σε ό,τι αφορά την ένταξη. Κυρία Κοπά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν θα επανέλθω σε θέματα που έχουν ήδη θέσει οι συνάδελφοι. Θέλω απλώς να πω ότι οι υποχρεώσεις από το πρωτόκολλο της Άγκυρας δεν μπορούν να παρακαμφθούν. Και σχολιάζοντας απλώς αυτό που είπε ο υπουργό ε, για μηδενικό προβλήματα με τους γείτονες, ε, συμφωνώ ότι τα ατμοσφαίριξ είναι πάντα καλά. Και η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Καραμαλή ήταν σίγουρα ένα θετικό σημείο στο γάμο ε, του παιδιού του κύριου Ερντογάν. Παρόλα αυτά θα ήταν πολύ καλύτερα και θα εξασφαλιζόταν πολύ ο στόχος των μηδενικών προβλημάτων αν η Τουρκία απέφευγε την διαρκή παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου και όλο το καλοκαίρι δεν προχωρούσε σε χαμηλές υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά, τρομοκρατώντας τους κατοίκους. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε από τα ατμοσφαίριξ και να έρθουμε στην ουσία. Κύριε Υπουργέ, μια συγκεκριμένη ερώτηση που θέλω να σας κάνω αφορά την έναρξη ε, των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Επανεισδοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών είναι ότι η Τουρκία θέλει να καθυστερήσει ακόμα την έναρξη των συζητήσεων. Θα ήθελα από εσά να επιβεβαιώσετε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καθυστέρηση στην έναρξη διαπραγματεύσεων. Και τέλος, να ρωτήσω αν, ε, ποια είναι η γνώμη σας για την εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα. Γνωρίζετε καλά ότι η Ελλάδα λαμβάνει από την Τουρκία 500 άτομα τη μέρα μέσω των θαλασσίων συνόρων. Ε, γι' αυτό η εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας που είχε υπογραφεί ανάμεσα στο σημερινό Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον αείμνηστο Τζέμ ε, χρειάζεται απαραίτητο να εφαρμοστεί. Ποια είναι η γνώμη σας. Ευχαριστώ. Κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Υπουργός απήντησε βέβαια σε διάφορα ζητήματα, αλλά επί της ουσίας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας και την μη αναγνώριση ενός κράτους μέλους που είναι η Κύπρος δεν απήντησε. Και το σημείο είναι χαρακτηριστικό. Είναι δυνατόν η Τουρκία να προχωρήσει στον ευρωπαϊκό δρόμο εάν δεν έχει εξασφαλιστεί και η καλή σχέση με τους γείτονες. Είδαμε το προηγούμενο της Κροατίας με τη Σλοβενία. Η Κροατία υποχρεώθηκε να συμφωνήσει σε ορισμένα πράγματα για να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προς την Ευρώπη. Πώς το αντιλαμβάνεται αυτό η τουρκική πολιτική τάξη. Επειδή ακριβώς σε ζητήματα που έχουν σχέση με το διεθνές στάτους ε, η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να μην ακολουθεί την ε, διπλωματική λογική που έχει επικρατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που δημιουργήθηκε. Αυτό θέλω να απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος Κατσίν. Ευχαριστώ κύριε Προβέρα. Αγαπητά κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ που ήρθατε εδώ και θα ήθελα να, συγχαρώ, να σας συγχαρώ για τον πολύ πιστικό σας λόγο, καθώς και για τις ε, αντιδράσεις που είχατε, ο Πρωθυπουργό σας κυρίως, για τα γεγονότα της ε, Γάζας. Διερωτώ με αν άλλοι πρωθυπουργοί θα μπορούσαν να είχαν αντιδράσει ε, τόσο στενάρα όπως ο πρωθυπουργό σας και να καταδικάσουν αυτά που έγιναν. Εκείνη την εποχή ο Πρωθυπουργό και η Τουρκία κέρδισαν πραγματικά μεγάλη έγκλη. Θα ήθελα λοιπόν γι' αυτό να σα συγχαρώ, ειλικρινά. Είπατε ότι χρειάζεται την υποστήριξή μα και την ενθάρρυνσή μα. Θα ήθελα να σα ενθαρρύνω να ολοκληρώσετε τη Συμφωνία Επανιστοχή. Γιατί αν χώρε που δεν είναι ακόμα υποψήφιε χώρε ε, στα Δυτικά Βαλκάνια αν αυτές οι χώρες μπορούν να συνάψουν συμφωνίε επανεισδοχή, τότε πολλό δε μάλλον μπορεί να το κάνει και η Τουρκία. Το Κωσυφοπαίδιο το έκανε. Ε, η Τουρκία μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο επίσης. Άκουσα τον λόγο σας και με βάση αυτό τον λόγο μπορούμε να εκτιμήσουμε το δυναμικό που έχει ε, η Τουρκία έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί δεν κάνει περισσότερα η Τουρκία. Είμαι πεπισμένο ότι μπορεί να κάνει περισσότερα και μπορεί να δουλέψει πολύ πιο ταχαίω. Θα ήθελα λοιπόν να σα ενθαρρύνω ε, το πρωτόκολλο το οποίο συμφωνήθηκε για να βελτιωθούν οι σχέσει με την Αρμενία να κυρωθεί από το κοινοβούλιο σα το συντομότερο δυνατόν. Η Τουρκία είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η επικύρωση από το κοινοβούλιο αυτού του πρωτοκόλλου θα αυξήσει την αξιοπιστία της Τουρκίας και στην περιοχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι από τα βασικά στοιχεία, τα βασικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να προοδεύσει περαιτέρω ε, στην ευρωπαϊκή της πορεία η Ευρώπη. Κάτι πιο συγκεκριμένο τώρα, μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Χρειάζεστε περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξή σας ε, συγκεκριμένα στα νότια-ανατολικά που είναι λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή. Μια άλλη επίσης ερώτηση. Είπατε ότι η ανακοίνωση για την επικοινωνία με το Ιράν δεν είναι ε, επαρκής. Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ε, τον κατάλληλο διάλογο με το Ιράν για να εμποδίσετε οποιαδήποτε πυρηνική εξέλιξη. Κύριος Μαυρονικόλας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην οποία ακούσαμε πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό δεν υπήρξε πιστική διότι ορισμένες από ενέργειες και πράξεις που έχουν γίνει έρχονται σε αντίθεση με τις πραγματικότητες. Μιλήσαμε για μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες, αλλά πιστεύω ότι η γενικότερη αντίληψη είναι ότι όλοι οι γείτονες πιστεύουν ότι έχουν προβλήματα με την Τουρκία. Αναφερόμενος στο κυπριακό πρόβλημα θα πω το εξής. Από το 2006 δεσμεύθηκε η Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας και να βοηθήσει στις συνομιλίες. Δεν έχει αναγνωρίσει ούτε την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία βλέπει μέσα από τις συνομιλίες λύση συνομοσπονδίας και όχι λύση ομοσπονδίας. Επίσης, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορεί κανείς με μεγάλη ακρίβεια να ισχυριστεί ότι από το 2006 και εντεύθεν η τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει σμικρινθεί σε αριθμόν. Σε αντίθεση, οι έπικοι έχουν αυξηθεί και σε ένα νησί με έναν εκατομμύριο πληθυσμών υπάρχουν αυτή τη στιγμή 400.000 έπικοι από την Τουρκία συν 40.000 τουρκικά στρατεύματα ετοιμοπόλεμα. Ανέμενε έμενε κανείς ότι η Τουρκία ως μεγάλη χώρα και μεγάλη δύναμη όπως ορθά ανέφερε ο κύριος Υφυπουργός θα μπορούσε να κάνει ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η Λευκοσία είναι μοιρασμένη πόλη και η Αμόχωστος πόλη φάντασμα. Μπορεί η Τουρκία να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ. Τσαβέλα, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Όταν είπαμε στον ε, κύριο Έλμαρ Μπρόκ ότι εσείς και εγώ είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια, μας ρώτησε ήσασταν φίλοι πριν γίνει επικίνδυνος ο κύριος ο κύριο Έγκεμεν Μπαγκή, υπονοώντα ότι τώρα που γίνατε υπουργό, μου είσαστε ένας επικίνδυνος φίλος. Κύριε Υπουργέ, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και οι δυο έχουμε δουλέψει πολύ επικοδομητικά για να βοηθήσουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να βρουν ένα μόντους λιβέντη. Ήμουνα προϊσταμένη Ελληνικού Ιδρύματος. Εδώ και δέκα χρόνια δίνουμε υποτροφίες σε Τούρκους φοιτητές για το Χάρβαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σας είχαμε και καλεσμένο πριν από δύο εβδομάδες, για να παρουσιάζετε σε ελληνικό ε, έδαφος, στο ελληνικό αυτό ίδρυμα, τις απόψεις της Τουρκίας. Κύριε Υπουργέ, καθαρά πράγματα γείτονες χώρες, πολιτική μηδενικών προβλημάτων με τους γειτόνους σας, κάζους μπέλη με την Ελλάδα. Γιατί, επί της ουσίας, επισύεται την απειλή να επιτεθείτε στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι επί της ουσίας. Νομοτελειακά και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, κάποια στιγμή η Ελλάδα θα είναι τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσείς εξακολουθείτε, γιατί το ξέρετε καλά, ότι γίνονται τουρκικές ενέργειες, και εδώ και πέντε χρόνια είχαμε σχεδόν και πόλεμο, από την Τουρκία προς την Ελλάδα, που οδηγεί την πατρίδα μου σε εξοπλισμού στην τελευταία πενταετία 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κύριε Υπουργέ, στερείτε τα χρήματα αυτά από τον ελληνικό λαό Στερείτε τα χρήματα αυτά από την παιδεία μας, την κοινωνική μας ασφάλιση. Κάζους μπέλι με την Ελλάδα. Τι θα κάνετε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαγκής για αυτά τα οποία είπε. Ωραία λόγια, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία έκφραση, δημοκρατία, αλλά δυστυχώς λίγα πράγματα στην πράξη. Πώς μπορείτε εσείς να έρχεστε σε επαφή και να είστε φίλοι με το Ιράν, με ένα τόσο αντιδημοκρατικό καθεστώς. Πώς μπορείτε να είστε μέλος του οργανισμού ε, της Ισλαμικής Διάσκεψης και να λέτε πως πρέπει να παραμείνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι εκεί που ορίζει η Σαρία και το έχει υπογράψει. Πώς μπορείτε όταν εγώ επισκέφθηκα τη χώρα σας να διώξετε τον τύπο. Επειδή άσκησε κριτική στο ρόλο της Τουρκίας στην Κύπρο. Το κάνατε εσείς κύριε Πρόεδρε μαζί με την κυρία Φλότρ. Σκάνδαλο. Και έδιωξε η δική μου πρόεδρος τον τύπο για να μην μιλήσω, να πω την άποψή μου για την Τουρκία. Πώς μπορεί ο πρόεδρος του κόμματός μου, ο Χέρτ Βίλτερς, που εκφράζει ελεύθερα την άποψή του και ασκεί κριτική για την ιδεολογία του Ισλάμ, πώς μπορείτε να του αρνείστε την είσοδο της χώρα, στην χώρα σας ως μέλος αντιπροσωπείας Ολλανδίας, του Κοινοβουλίου. Πώς τολμάτε να μιλάτε για ελευθερία γνώμης, για την κατοχή, την κατοχή την παράνομη της Κύπρου. Πρέπει το 2010 να φύγουν τα στρατεύματά σας από την Κύπρο. Κατέχετε παράνομα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό συμφωνούμε όλοι εδώ μέσα. Κατόπιν, τι είπατε για το δημοψήφισμα της ε, Κύπρου και για το, με συγχωρείτε, για το δημοψήφισμα το πρόσφατο για το ότι δεν επιτρέπεται να χτίζουν πλέον ε, μιναρέδες στην ε, Ελβετία. Σκεφτείτε τι κάνετε στους χριστιανούς στην Τουρκία. Κατόπιν, κάποιοι λόγοι για τους ε, οποίους θεωρούμε πως δεν πρέπει να γίνει η Τουρκία ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να το συζητήσουμε δεν έχουμε χρόνο, αλλά αυτή είναι η άποψή μας. Υπάρχουν λόγοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ, να συγχαρώ την Τουρκία για δύο πράγματα εξίσου ε, εξόχω σημαντικά που συνέβησαν μέσα στο 2009. Καταρχάς, για τη συμφωνία Ναμπόκο, νομίζω ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι είναι ικανοποιημένοι για την ε, υπογραφή αυτής της συμφωνίας και δεύτερον, για την συμφιλίωση με την Αρμενία. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ. Όμως, όπως ε, υπόθηκε κατ' επανάληψη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Τουρκία ε, σημειώνει πολλές καθυστερήσεις ό,τι αφορά τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Η ερώτησή μου θα είναι λοιπόν πολύ ευθεία. Βασίζομαι σε κάποια αριθμητικά στοιχεία. Είδα ότι το 2002 74% των Τούρκων ήταν υπέρ της ένταξής σας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως το 2009 μόνο το 45% των Τούρκων είναι υπέρ της ένταξής σας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει σχέση μεταξύ της μείωσης του ενθουσιασμού και τις ε, βραδιπορίες με την οποία σημειώνεται τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκζίμη. E, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι όπως και σας άκουσα με, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή την ομιλία σας όπου μας παρουσιάσατε όλα τα επιτεύγματα της Τουρκίας τα εσωτερικά, τα πολιτικά και την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Ξέρω ότι είναι μια δυσχερής διαδικασία και ήταν πολύ σπουδαία εμπειρία και για την Πολωνία όταν ε, είχε τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις. Θα περιμέναμε να ήταν πιο εύκολα ορισμένα κεφάλαια για την Τουρκία σε ό,τι αφορά τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις. Άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον για το Ιράν. Είπατε ότι η Ανατολική Ευρώπη καταλαβαίνει καλύτερα το Ιράν από ό,τι Κεντρική Ευρώπη ή Δυτική Ευρώπη. Μήπως θα μπορούσατε, θα είχατε την καλοσύνη να αναλύσετε τι ακριβώς εννοείτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκθεση που μας παρουσίασε το πρωί η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Και τις εκτιμήσεις ε, από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία συμμετείχε και ο πρέσβης της χώρας σας. Είχαμε πολλές ε, επιφυλάξεις μη κυβερνητικών οργανώσεων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των διατάξεων ε, για, κατά της τρομοκρατίας και ιδιαίτερα του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων που θεωρούν πολύ δύσκολη τη θέση της, πώς ε, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε αυτά τα θέματα του άρθρου 301 του ποινικού κώδικα. Ο κύριος Αλαβράκος. Κύριε Υπουργέ, είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Τουρκία, όπως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τις Ηνωμένε Πολιτείες, χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία και όλα τα κράτη τα οποία απαρτίζουν τη διεθνή κοινότητα. Ελπίζω αυτό να το θεωρείτε κι εσείς ότι είναι σωστό. Επίσης, εκείνο το οποίο θέλω να σας πω ότι αντελήφθην τον υπενιγμό σας ότι 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι μου στην κοινότητα α, προσδοκούν με αγωνία τα αποτελέσματα αυτής της συναντήσεως και της εν γέννη εξελίξεως της υποθεσεώς σας. Θέλω να πω όμως και να σας υπενθυμίσω ότι το μεταναστευτικό συνάλλαγμα είναι ένας βασικός πόρος με τον οποίο σώζεται η χώρα σας οικονομικά. Και αυτό οπωσδήποτε φιλείται στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Τώρα, θέλω να επισημάνω τα εξή. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσία στη χώρα σας, τα οποία το ένα με το άλλο αντιπαρατίθενται. Και αυτά τα κέντρα εξουσία κατά βάση είναι η κυβέρνηση που αποτελεί τη λαϊκή κυριαρχία. Το δεύτερο είναι ο στρατό, ο οποίο έχει δική του πολιτική. Και το τρίτο είναι η δικαιοσύνη. Ήδη μέσα στον χρόνο είχατε πρόβλημα επαναλήψεως του φαινομένου της κυβερνήσεως Ερμπακάν. Το δεύτερο είναι ότι ο στρατός τη στιγμή που εσείς χαμογελάτε προς την Ελλάδα κάνει συνεχείς παραβιάσεις των ελληνικών συνόρων με υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Και το τρίτο είναι ότι η κυβέρνησή σας αυτή τη στιγμή δεν δίνει σαφή σημεία από το οποίο να προκύπτει ότι μπορεί να αντιθασεύσει τα άλλα κέντρα εξουσίας και να τους δημιουργήσει την εντύπωση ότι η λαϊκή κυριαρχία στη χώρα σας είναι βασική πηγή εξουσίας. Από την άλλη πλευρά, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι προσφάτως το Σεράγεβο επεδείχθη μια τάση συγγυμονεύσεως με την δημιουργία ενός είδους κοινοπολιτείας κατά τα πρότυπα της Βρετανικής κοινοπολιτείας. Ποια τελικά είναι η άποψή σας. Είσαστε μέσα στο πνεύμα της συνθήκης της Ρώμης του άρθρου 49 το οποίο αποτελεί την πηγή της συνθήκης και των ορίων της Κοπενχάγης ή δεν είστε. Προτελευταίος ομιλητής, η κυρία προτελευταιος ομιλητη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να θέσω μια ερώτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί συχνά το συζητάμε σε πολλές εκθέσεις ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερία του τύπου, έκφρασης, αλλά έχω την αίσθηση πως ε, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται είναι ένα άρθρο από εδώ, ένα άρθρο αφαιρείται, προστίθεται. Δεν είναι δηλαδή μια ενιαία πολιτική ελευθερίας ε, του τύπου. Και ξανά επανέρχεται το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Το ίδιο ισχύει παραδείγματος χάρη και για τη θρησκευτική ελευθερία. Νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό ζήτημα για ολόκληρη την Ευρώπη και για την ε, Τουρκία. Βλέπετε πως αυξάνεται η μη ανεκτικότητα όσον αφορά τις άλλες θρησκείες. Οπότε θέμε η Τουρκία να έχει σωστή θέση. Δεν μιλάω μόνο για τις ε, χριστιανικές μειονότητες, για όλες τις ομάδες. Έχουμε δηλαδή έτσι εμβαλωματικές ε, λύσεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα ενιαίο όραμα το οποίο θα εφαρμόσετε και νομίζω πως θα πρέπει είτε να αλλάξει το σύνταγμα είτε να συνταχθεί ένα νέο σύνταγμα. Αυτό είναι ο ιδεώδης τρόπος. Σκοπεύετε να αναλάβετε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ποιες είναι οι ιδέες σας ε, για να λυθούν αυτά τα ζητήματα άπαξ και διαπαντός. E- Ο κύριος Αγκουράκης και συνεχεία λίγιο χρόνος. Παρακαλώ. Το ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα δύο τις επισημάνσεις στις παρεμβάσεις του κυρίου Υπουργού. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, είχα διαβάσει για τον ε, νεοοθωμανισμό που εμφανίζεται στην Τουρκία. Δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αλλά πρέπει να πω ότι η παρεμβάση του κύριου Υπουργού, οι δύο σήμερα, ε, ήταν άκουσα αποκαλυπτικές για μένα και πρέπει να ανησυχήσω. Το δεύτερο που ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό είναι ότι χαίρομαι ιδιαίτερος για τα μέτρα προόδου στην Τουρκία. Θεωρώ όμως ότι τα μέτρα αυτά είναι περισσότερο ζητήματα ορίμανσης του εργατικού και προοδευτικού κινήματος στην Τουρκία και όχι κάποιο δώρο ε, της κυβέρνησης που έχει την τιμή να εκπροσωπεί εδώ. Και με την έννοια αυτή να πω ότι δεν θεωρώ για κάτι πολύ σπουδαίο μετά από 50 χρόνια να αποδοθεί η ηθαγένεια στον πολύ μεγάλο Ναζίμ Χικμέτ και να μας το παρουσιάζει ο κ. Υπουργό ως μεγάλο επίτευγμα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και παγκόσμια κουλτούρα. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι καλές είναι οι επενδύσεις και 20 ε, φορές παραπάνω ξένες επενδύσεις στην Τουρκία αλλά δεν μας είπε τίποτα για, την, ε, για το μεγάλωμα της ψαλίδας μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων που ειδικά στη χώρα του είναι πάρα πολύ έντονο και έτσι ε, εξηγούνται και διάφορες κοινωνικές εκρήξεις που υπάρχουν εκεί. Τέλος, θα ήθελα το εξής, το, ε, ε, το 301 του κωδικού νόμου, του ποινικού κώδικα, αν δεν με απατάει η αφορά, ε, πρόσβαση, αφορά ύβρις προς το τουρκικό κράτος. Αν αυτό το πράγμα διατηρείται, δεν μπορείτε κύριε Υπουργέ να μιλάτε για τα δικαιώματα των Κούρδων. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω το εξή: Εάν συνεχίσετε με τις υπερπτήσεις των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, είναι γνωστά τα επιχειρήματά σας, αναρωτιέμαι πότε θα έρθει η στιγμή να βλέπουμε τα τουρκικά αεροπλάνα και πάνω από την Αθήνα, διότι έτσι πως πάει, δεν φαίνεται να αναγνωρίζετε σύνορα στον αέριο χώρο τουλάχιστον του Αιγαίου. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Τελευταίος, ο κύριος Τάνοκ για το ζήτημα της ε, Τουρκίας και τον ρόλο της εντός του οργανισμού της Ισλαμικής Διάσκεψης. Ε, να δούμε λίγο πού πιθανώς έχουμε συγκρούσει στο μέλλον για τις αξίες που αναφέρατε. Μιλήσατε για την διακήρυξη του Καΐρου, αλλά αυτό το οποίο μας ανισχύει είναι πως είχατε προσκαλέσει την ηγεσία της Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση δηλαδή, ε, στην Άγκυρα και ε, ενώ είχατε προσκαλέσει τον πρόεδρο Μπασίρ σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, ε, αναζητείτε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αν και τελευταία στιγμή δεν ήρθε μετά από διεθνή πίεση. Οπότε πρέπει να το δει αυτό η κυβέρνησή σας πολύ προσεκτικά. Επίσης, θίξατε το ζήτημα πως ε, υπάρχει είναι ισοδύναμη η παρουσία των κυρίαρχων βάσεων με τα δικά στρατεύματα. Να σα υπενθυμίσω ότι η Συμφωνία Εγγύηση του 1960 δεν έχουν ούτε μία σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία οι κυρίαρχε βάσει. Είναι κυρίαρχο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και όλε οι πλευρέ συμφωνούσαν με την παρουσία μα. Δεν τίθεται ζήτημα. Αν και μέρο τη επικράτεια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τη Βρετανική κυβέρνηση θα επιστραφεί ω επιπράβευση τυχόν συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Επίση, στα σχόλιά σα για την Αρμενία, ο συνάδελφο από του Εργατικού μίλησε για πρόοδες, μιλήσατε για πολλέ δυνατότητε. Ω φίλο τη Αρμενία, απογοητεύομαι λίγο. Μετά από όλο το πολιτικό κεφάλαιο που επένδυσε ο πρόεδρο Σαρκοζή στο να μεταπίσει τη διασπορά, την επομένη νομίζω είπε ο Πρωθυπουργό σα πω εάν ε, δεν λυθεί η διαμάχη νομίζω, του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν θα ανοίξουν τα σύνορα. Βεβαίως πράγματι υπάρχει διαμάχη με το Αζερβαϊτζάν, αλλά πώ ε, εξηγείται το ότι το Καζακστάν, μια άλλη τουρκογενής χώρα, έχει σχέσεις χωρίς να του εμποδίζει αυτό. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσετε το ζήτημα του Αζερβαϊτζάν και να περάσετε σε μια συμφιλίωση. Thank you. Και ο Ευχαριστώ. Ήξερα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεγάλο θεσμό, αλλά σήμερα το αισθάνθηκα στα κοκαλά μου, στη σάρκα μου. Με όλε αυτέ τι ερωτήσει, με όλο αυτό το ενδιαφέρον που έχει η Τουρκία, ε, κάτι που με γεμίζει με υπερηφάνεια. Ε, έχω το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο τελικά. Ε, όλες αυτές οι ερωτήσεις, όλες αυτές οι επικρίσεις ε, με κάνουν να αισθάνομαι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τελικά είναι σημαντικό. Το να φέρουμε δηλαδή την Ευρώπη και την Τουρκία κοντά. Σε ό,τι αφορά τις διστάμενες απόψεις που ανέφερε ο κύριος Σαλαφράνκα από διάφορους ε, ηγέτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς επηρεάζει τους ε, Τούρκους πολίτες. Σε μια σφιγμομέτρηση φάνηκε ότι 60% των Τούρκων επιθυμούν οι Τούρκοι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν τους ρωτήσαμε, πιστεύω ότι θα μπει η Τουρκία, το 40% είπε ναι και η διαφορά του 20% έχει να κάνει με την έλλειψη εμπιστοσύνη που προκύπτει από κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει. Αλλά όλοι πολιτικοί είμαστε στο κάτω-κάτω και σε κάποιες χρονικές στιγμές χρειάζεται να κάνουμε κάποιες δηλώσεις ανάλογα με το πολιτικό αέρα ε, και κύμα που φυσάει. Αλλά τελικά ξέρετε ότι αυτό που προσπαθούμε κι εσείς κι εμείς ε, είναι πολύ σωστό εκπολιτιστικό καθήκον το να έρθει κοντά η Τουρκία στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό ε, και για τους δυο μας αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Για τα, τις ερωτήσεις κυρία Σκοπά, για τις διαφορές ε, απόψε μεταξύ Τουρκίας και Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργό μου είχε μια μακρά συνομιλία ε, με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη μια εβδομάδα μετά τις ελληνικές εκλογές. Εγώ επισκέφθηκα την Αθήνα και ο Πρωθυπουργό μου έστειλε μια επιστολή τετρασέλιδη επιστολή στον Πρωθυπουργό Παπανδρέου, όπου τον ρωτούσε αν μπορεί να συνεργαστεί για θέματα μειονοτήτων και στις δύο χώρες, για το θέμα της Κύπρου, για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και για το θέμα της λαθομετανάστευσης. Στο τέλος της επιστολής μου, ο Πρωθυπουργό προσφέρθηκε να συνεργαστούν ε, τα Υπουργικά Συμβούλια υπό την αιγίδα των δύο Πρωθυπουργών για να ε, συζητήσουν για τα θέματα που μας ενώνουν και μας διαιρούν. Και περίμενε την απάντηση του κύριου Παπανδρέου, αλλά όταν τον ε, συνάντησα δύο μέρες μετά, είχε λάβει την επιστολή που ήταν πολύ θετική η απάντηση. Είμαι λοιπόν και εγώ αισιόδοξο. Υπάρχουν ε, διαφορέ, αλλά σε σχέση με το παρελθόν μα με το παρελθόν μας είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε διερευνητικέ συζητήσει για το Αιγαίο για να θέσουμε τέρμα σε αυτές τις διαφορές. Για το πού ξεκινάνε τα εναέρια σύνορα, ε, για τις ερμηνείες μας που μπορεί να είναι διαφορετικές. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να έχουμε ηγέτες με θάρρος, με τόλμη, που θα συνεργαστούν, που θα συνομιλήσουν και που θα σφίξουν ένα στο χέρι του άλλου. Δεν υπάρχει καθυστέρηση από πλευρά Τουρκία για την Συμφωνία Επανιστοχή. Είχαμε προγραμματίσει να οργανώσουμε τη συνάντηση στις 4 Δεκεμβρίου στην Τουρκία με τον Γενικό Διευθυντή. Αλλά επειδή αλλάζουν τα χαρτοφυλάκια στην Κομισιόν και επειδή ο Γενικός ε, Γραμματέας, ε, Διευθυντής αυτός αναλαμβάνει νέο χαρτοφυλάκιο, θα αναβάλουμε τη συνάντηση. Αλλά μόλις ε, θα εγκριθεί το νέο σώμα των Επιτρόπων, και θα αναλάβουν τα νέα πρόσωπα, θα συνεχίσουμε. Θέλουμε να επιλύθει αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι ελληνοτουρκικό θέμα. Είναι ευρωπαϊκό θέμα και η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Για το θέμα της Κύπρου. Σέβομαι τις προσδοκίες και τις απόψεις όλων των εκπροσώπων της, της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτήν την αίθουσα. Αλλά θα πρέπει και οι δύο να καταβάλουμε προσπάθειες. Αν είχε περάσει το δημοψήφισμα, θα ήμασταν σε μια τελείω διαφορετική κατάσταση σήμερα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Η θέση της Τουρκίας βασίζεται στα όσα λέει ο ΙΕ. Μια συνολική λύση, το συντομότερο δυνατόν, που να βασίζεται στη διζωνική, δικοινοτική λύση. Με ισότητα. Δεν μιλάμε για ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Δεν χρησιμοποιούμε τέτοιες ε, ε, εκφράσεις. Όσο υπάρχει πολιτική ισότητα όσο ε, οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι αισθάνονται άνετα με αυτή τη λύση ε, για το μέλλον τους, θα τους υποστηρίξουμε. Και θα σας πω ειλικρινά το εξή. Αν εγώ ήμουν Κύπριος, Έλληνας ή Τούρκος Κύπριος, εγώ θα ήμουν υπέρ της ε, ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η ένταξη της Τουρκίας για την Κύπρο και για όλη την περιοχή να συνεχιστούν αυτέ οι διαπραγματεύσει. Ελπίζω αυτό το θέμα να μα ε, συνενώσει και θα συνεργαστούμε για αυτό το περαιτέρω. Τώρα, για τη συμφωνία επανεισδοχή, θα ήθελα να πω. Θέλουμε να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό εφόσον υπάρχει επιμερισμό των βαρών. Ε, δυσκολευόμαστε και εμεί να εξηγήσουμε στο λαό μα ότι ω μέλο τη Τελωνιακή Ένωση, ε, τη στιγμή που τα αγαθά μα κινούνται ελεύθερα στον ευρωπαϊκό χώρο οι ιδιοκτήτε αυτών των αγαθών πώ γίνεται να μην μπορούν. Δεν έχει νόημα. Επομένω θα πρέπει να σταματήσουμε ε, με αυτό το φραγμό ας πούμε, των θεωρήσεων για του πολίτε τη Τουρκία. Γι' αυτό όμω, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να επιληθεί το κόλλημα τη Συμφωνία Επανεισδοχή. Γι' αυτό θα θέλαμε να δούμε μία λύση σε αυτό το θέμα. Το συντομότερο δυνατόν. Για το αν χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για την Ανατολική Τουρκία. Εμεί ήδη διοχετεύουμε ε, κονδύλια ε, προς αυτήν την κατεύθυνση. Φέτος δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ. Ε, θα, τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα δοθούν περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί θέλουμε να υπάρξει πρόοδος ε, και στι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχές της Τουρκίας. Το γεγονό ότι το κόμμα μου έλαβε 25% των ψήφων σε αυτή την περιοχή το 2002 και 60% των ψήφων το 2007, αυτή η διαφορά δείχνει πραγματικά ότι ο λαό τη περιοχή καταλαβαίνει ότι ενδιαφερόμαστε για τα προβλήματά του και ότι είμαστε αποφασισμένοι να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Τώρα, υπάρχει αντίφαση. Ε, στις σχέσεις μας με τους ε, γειτονές μας. Η πρόθεσή μας είναι να μην υπάρχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να, και αυτοί να κάνουν προσπάθεια. Θέλουν να επιληθούν τα προβλήματα εφόσον υπάρχουν εταίροι ε, πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας με τη Συρία. Ε, το γεγονός ότι έχουμε καλύτερες σχέσεις με το Ιράν, ότι έχουμε καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία, ε, με τη Βουλγαρία, με τη Ρουμανία, με τη Γεωργία. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε να επιλύσουμε επίση και τα προβλήματα και με του υπόλοιπου γείτονε. Και είμαστε αποφασισμένοι να προσπαθήσουμε. Έχουμε 13 γείτονε, 13 όμορε χώρε. Καμία χώρα δεν επιλέγει τους γειτονές της φυσικά. Και οι γείτονες μας δεν είναι εύκολοι γείτονες. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με αυτούς. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι για το κοινό καλό κάτι τέτοιο. Για το κάσους Μπέλη που υπάρχει ε, και το θέμα του διαλόγου. Νίκη, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Οι δύο ε, πρωθυπουργοί θα πρέπει να ενθαρρυνθούν. Η... Το κόμμα σα είναι στην αντιπολίτευση και θα πρέπει να υποστηρίξει τον κύριο Παπανδρέου και να τον ενθαρρύνει για να συζητήσουμε για αυτά τα δύσκολα ε, θέματα με του Τούρκου ομολόγου του. Αυτά τα θέματα μπορούν να λυθούν μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφού καταλάβουμε ο ένας τον άλλο. Έχουμε την θέληση για να τα επιλύσουμε. Μπορούμε να τα επιλύσουμε για τα ερώτηματα του κ. Μάλτνερ. Ο κ. Βίλτερ. Ε, μπορεί να μιλήσει ελεύθερα και να πει την άποψή του, όπως θέλει. Και εγώ επίσης μπορώ να πω τη δική μου α, άποψη, αλλά μπορώ και να μην ακούσω αυτά που λέει. Μπορώ να, μπορεί να μιλήσει, μπορεί να πει τα δικά του και εγώ τα δικά μου. Ο πρωθυπουργός σα, ο Ολλανδός πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι οι τουρκικές αρχές δεν χρειάζεται καν να τον συναντήσουν όταν πηγαίνει στην Τουρκία. κύριος Βίλτερς, ε, μερικές φορές είναι επικριτικός και χιδαίος. Ε, πριν να κρίνει τις αντιδράσεις των άλλων, να ακούσει αυτά που λέει ο ίδιος Ποτέ δεν ζητήσαμε από τους δημοσιογράφους να φύγουν από την ε, αίθουσα. Οι εισαγωγικοί λόγοι ε, στις κοινέ ε, κοινοβουλευτικές συναντήσεις θα πρέπει να είναι ανοιχτές στον τύπο και αυτό ανακοινώνεται, και αυτό ανακοινώνεται εκ των προτέρων. μετά από τις παρεμβάσεις, τις εισαγωγικές στην άγκυρα της κοινή Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, όπου η τουρκική πλευρά παρέθεσε τις απόψεις και εν συνεχεία η ευρωπαϊκή πλευρά τις δικές της. Ακόμη και ο πρόεδρος της τουρκικής ε, εθνοσυνέλευσης μίλησε και εγώ μίλησα και μόνο μετά έφυγε ο τύπος. Εν συνεχεία ενημερώσαμε τα μέλη του τύπου, επομένως τίποτα δεν παρέμεινε αδιαφανές και μυστικό. Είναι μια συνήθις διαδικασία αυτή. Για τους ε, μιναρέδες, οι χριστιανοί έχουν το δικαίωμα να χτίζουν τις εκκλησίες τους στην Τουρκία. Ναι, φυσικά έχουν αυτό το προνόμιο εδώ και 800 χρόνια. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν ε, συναγωγές, ε, τζαμιά και εκκλησίες δίπλα-δίπλα. Εγώ ζω σε μια γειτονιά, σε μια πολυκατοικία, όπου τα παιδιά μου παίζουν με βρεόπουλα και χριστιανόπουλα. Και τα παιδιά μου παίρνουν δώρα ε, όταν υπάρχει οποιαδήποτε θρησκευτική οργή, ε, γιορτή εβραϊκή, χριστιανική κτλ. Γιορτάζουμε τις, ε, όλες τις θρησκευτικές γιορτές. Είναι ένας χώρος όπου συνεπάρχουν όλα. Φυσικά αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, αλλά τα τελευταία 800 χρόνια αποδείξαμε ότι οι διαφορετικές κουλτούρες, οι διαφορετικές θρησκείες, οι διαφορετικές γλώσσες, οι διαφορετικές εθνότητες μπορούν να συνεπάρξουν. Και πιστεύουμε ότι αυτό πλουτίζει την Τουρκία. Και ελπίζω ότι η κυβέρνηση της Ελβετίας δεν θα θέσει τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε δημοψήφισμα σε μικρές πόλεις. Αν η Ελβετία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έκανε τέτοια πράγματα. Δεν θα ψηφιζόταν εκεί αυτά τα θέματα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξασφαλίζει μόνο την ευημερία των μουσουλμάνων στην Ευρώπη, αλλά και την ευημερία των χριστιανών, των Εβραίων, των άθεων σε οποιοδήποτε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, όπως σας είπα, είναι το μεγαλύτερο ενευτικό project της παγκόσμιας ε, ιστορίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον Αμπούκο. Σήμερα το πρωί είχα μια συνάντηση με τον σημερινό Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Πιμπάλξ, και η Τουρκία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει αυτή την ε, πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι το Ναμπούκο είναι ένα ε, έργο που το χρειαζόμαστε και η Τουρκία θα εξακολουθήσει να είναι τμήμα του κάθε της λύσης του κάθε ευρωπαϊκού προβλήματος, καθώς και της ενέργειας. Θα ήθελα Επίσης θα ήθελα ε, για το θέμα του αγωγού να υπάρχουν πολλές διαφορετικές πηγές, οδοί, μεταφοράς του κτλ. Για το Ιράν. Όταν μίλησα για την Ανατολική Ευρώπη εννοούσα την ε, Τουρκία. Γιατί εμείς είμαστε ε, μια ευρωπαϊκή χώρα στα ανατολικά της Υπήρου. Έχουμε σύνορα όμως με, με το Ιράν. Και χάρη σε αυτή την εγκύτητα έχουμε μάθει να επικοινωνούμε με το Ιράν το 1 τρίτο των Ιρανών, το πιστεύετε ή όχι, μιλούν τουρκικά και μάλιστα θαυμάσια. Ε, έχουμε καλύτερα επικοινωνιακά ταλέντα και προσόντα από ό,τι άλλες χώρες. Ε, μη θεωρήσετε ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να απομονώσουμε έτσι, γεωγραφικά τη χώρα μας. Όχι, είμαστε εναντίον όλων των διαφορών, όλων των εμποδίων και διακρίσεων και οι λύσεις θα πρέπει να είναι κοινέ. Μην ξεχνάτε ότι οι Ιρανοί είναι πολύ πεπειραμένοι διπλωμάτες. Τα δύο έθνη σε αυτό το τμήμα του πλανήτη που είχαν κράτη δικά τους πάνω από χίλια ε, χρόνια ήταν οι Τούρκοι και οι Πέρσες. Ε, Επικοινωνούμε λοιπόν μαζί τους και τους ενθαρρύνουμε να επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο, με την ε, Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Έχουμε εμπόριο με αυτούς και οι περισσότερες από τις χώρες έχουν πολύ περισσότερες εμπορικές ανταλλαγές ε, με το Ιράν από εμάς. Ε, ελευθερία του τύπου, θεμελιώδη δικαιώματα. Όλα αυτά τα πράγματα βελτιώνται στην Τουρκία. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχουμε επιλύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά για την ελευθεροτυπία ομολογώ ότι τα τελευταία 7 χρόνια δεν πέρασε ούτε ένα νομοθέτημα από, το, από την τουρκική εθνοσυνέλευση για να μειωθεί η ελευθερία του λόγου ή η ελευθερία των ημιέψιλων. Έχουμε χιλιάδες νόμους για να εξασφαλίσουμε την ελευθερία του τύπου. Υπάρχει ένα φορολογικό θέμα ε, που επέβαλε, ένας φόρος που επέβαλε η εφορία και το Υπουργείο Οικονομικών σε έναν όμιλο ΜΜΕ. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη ούτως ή άλλως αρχή που αποφάσισε για το φόρο. Αν το είχε ε, αποφασίσει να επιβάλλει, να φορολογήσει μια τράπεζα, δεν θα είχε θεωρηθεί ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε τις τραπεζικές συναλλαγές. Παντού, ε, σε κάθε χώρα, ε, ο καθένας πρέπει να πληρώνει του φόρους του και στην Τουρκία. Αυτή η εταιρεία, αυτός ο όμιλος, είχε προβλήματα με, την εφορία μας στο παρελθόν και αποφάσισε να υπάρξει διακανονισμός. Συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι συνομιλίες. Αν σταματήσουν τις συνομιλίες μπορούν να πάνε στα ανεξάρτητο δικαστήρια. Τα δικαστήρια της Τουρκίας είναι τόσο ανεξάρτητα ε, σε απόλυτο βαθμό. Το 85% των εταιρείων που αποφασίσουν να μην ρυθμίσουν τα φορολογικά τους, αλλά να πάνε ε, στο δικαστήριο, κερδίζουν τις αγωγές τους. Και αυτό δείχνει τις δραστηριότητες αυτού του δικαστηρίου. Αυτές οι εταιρείε που αποφασίζουν να μην προβούν σε διακανονισμό, μπορούν να προσφύγουν λοιπόν στον εξάρτητο δικαστήριο για φορολογικά θέματα. για το νέο Οθωμανισμό και το ερώτημα αυτό που έγινε, υπάρχει μια, ένα πρόβλημα ερμηνείας. Δεν έχουμε καθόλου τέτοιες ε, φιλοδοξίες. Απλώς έχουμε νέα, μια νέα προοπτική ως ε, δημοκρατία της Τουρκίας. Ε, και αυτό είναι η οικοδόμηση της ειρήνης. Γι' αυτό ακριβώς μεσολαβούμε, διαμεσολαβούμε σε όλες αυτές τις χώρες. Γι' αυτό εκλεγήκαμε για να εκπροσωπηθούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, του, ΟΗΕ μετά από 47 χρόνια. Και 8 από τα 10 κράτη του κόσμου ε, ψήφισαν την Τουρκία. Να είναι παρούσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο κύριος Μπασίρ δεν εκλήθη από την τουρκική κυβέρνηση. Στην Τουρκία τον κάλεσε η γραμματεία της Ισλαμικής Διάσκεψης για μία σύνοδο κορυφής ενός διεθνούς οργανισμού ε, που η χώρα του είναι μέλος. Δεν αποφασίζουμε εμείς ποιος θα προσκληθεί στην Ισλαμική διάσκεψη. Αυτό το κάνει η γραμματεία της ε, Ισλαμικής διάσκεψης. Καλεί τους αρχηγούς ε, κρατών κυβερνήσεων. Και αυτός επέλεξε να μην έρθει. Όσον αφορά τις κυρίαρχες βάσεις στην Κύπρο. Οι ίδιες εγγυήσει επιτρέπουν και σε εμάς, στην Τουρκία, να διατηρούμε στρατεύματα εκεί. Στην ίδια μοίρα είμαστε. Εάν είναι να το συζητήσουμε όμως πρέπει να μιλήσουμε τους πρόεδρους ε, Ταλάτ και Χριστόφια. Τώρα, γιατί να μην παραμερίσει τη σχέση της με το Αζερβαϊτζάν η Τουρκία όπως κάνει το Καζακστάν και έχει σχέση με την Αρμενία. Η Τουρκία επέδειξε την καλή της θέληση με το να υπογράψει το πρωτόκολλο. Και θα θέλαμε να κυρωθεί και από το Κοινοβούλιο. Αλλά πέραν κάποιων πολιτισμικών ομοιοτήτων, ε, γλώσσας και γειτονίας με το Αζερβαϊτζάν, έχουμε και 30% του αερίου που εισάγουμε από το Αζερβαϊτζάν πολλοί σύμμαχοι Ευρωπαίοι περιμένουν η Τουρκία να προωθήσει τον Ναμπούκο και η χώρα που θα το προμηθεύει το αέριο είναι το Αζερβαϊτζάν. Ε, ε, φάσκεται και αντιφάσκεται. Θέλετε η Τουρκία να μην να χαλάσει σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν. Εμείς θέλουμε πρόοδο, να δούμε πρόοδο και στις σχέσεις Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας όσον αφορά το Καραμπάχ, που θα είναι κάτι το υποφελές για όλο τον Νότιο Κάυκασο και η Γεωργία. Θα υποφεληθεί η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρωσία, η Τουρκία και θα έχουμε περισσότερη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή ολόκληρη. Παρακαλώ συνεχίστε να μας ε, στηρίζετε Ρία με την έκθεσή σας το πρώτο σχέδιο οπωσδήποτε θα εμπλουτιστεί, με σίγουρος, με από μέλη της Επιτροπής. Οι ιδέες σας, οι προτάσεις σας, οι απόψεις σας είναι πολύ σημαντικές για εμάς, γιατί είστε οι αιρετοί εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Οι συνεισφορές σας εκτιμώνται στην Τουρκία και να είστε σίγουροι πως είστε όλοι ευπρόσδεκτοι και να έρθετε και να ασκήσετε κριτική όσον αφορά το πώς θα έρθει πιο κοντά η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2010 είναι κρίσιμο έτος. Στη χώρα μας δεν έχουμε εκλογές. Στην Ευρώπη θα μετασχηματίσετε την Ένωση με μια νέα επιτροπή, με μια νέα συνθήκη με νέους κανόνες. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν το 2010 για να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει για τους ψηφοφόρους μας που είμαστε περήφανοι που τους εκπροσωπούμε και να κάνουμε τον κόσμο ασφαλέστερο και καλύτερο. Όχι για εμάς αλλά και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπάγκη για την παρουσία του, για τι παρεμβάσει του. Ελπίζω να τον ξαναδούμε σύντομα με καλά νέα και για την Τουρκία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα καλά νέα. Σα ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε εκ νέου. Έχουμε τον κύριο Μιγκαρέλη μαζί μας, τον κύριο Ιγκ Μιγκαρέλη, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα μας μιλήσει για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία. Και επομένως, θα μας εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση σήμερα και ποιες είναι οι πιθανές εξελίξεις. Τον καλωσορίζω λοιπόν. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί υπάρχει αυτή η αναβολή. Το Συμβούλιο τον περασμένο μήνα αποφάσισε να επεκτείνει κατά ένα χρόνο ε, την αναστολή στις ελευθερίες κίνησης ε, πολιτών της Λευκορωσίας. Και να, κάνει, να στείλει μηνύματα για διάλογο για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Επίσης, το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την ε, συμμετοχή της Λευκορωσίας στην εταιρική σχέση της ε, ανατολικής γειτονίας Κάτι πολύ σημαντικό που ενδιαφέρει έξι ανατολικέ χώρες, μεταξύ των οποίων και η Λευκορωσία. Θα θέλαμε να εκφράσουμε μια θετική στάση, ε, στηρίζουμε κάτι τέτοιο. Ε, εξάλλου, τα διάφορα ψηφίσματα μαρτυρούν ακριβώς αυτό. Είναι σημαντικό βαθμία να δημιουργήσουμε ένα διάλογο και θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα ε, από πλευρά Λευκορωσία ό,τι αφορά τι ατομικέ ελευθερίε, τον εκλογικό νόμο κτλ. Ο διάλογος αυτός σε καμία περίπτωση θα πρέπει να θέτει ένα αμφιβόλο τις επαφές με την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Επομένω, με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε όσα έχει να μα πει ο κ. Μιγκαρέλη για, την εξε... για τι εξελίξει των σχέσεων και τι διαπραγματεύσει για την σύναψη μια συμφωνία με τη χώρα αυτή. Κύριε Μιγκαρέλη, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας περιγράψω συντομία τη θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη Λευκορωσία. Και να σας πω ποιες ήταν οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Λευκορωσία. Χάρη ενός μεγαλύτερου εκδημοκρατισμού που θα πρέπει να συνεχιστεί και να εδραιωθεί στη χώρα αυτή. Ποια είναι λοιπόν η ανάλυση μας αυτή τη στιγμή. Όπως θα ξέρετε, από το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πολύ στενές σχέσεις με τη Λευκορωσία, γιατί το 1997, μετά την ανάληψη της εξουσίας ή μάλλον την εκλογή του πρόεδρου Λουκασέγκο και των περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν στη χώρα αυτή, το Συμβούλιο αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ε, υπογραφή και κύρωση της ε, Συμφωνίας εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας που είχε διαπραγματευτεί με τη χώρα αυτή, όπως και με όλες τις ε, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κατά το πρώτο ήμιση της δεκαετίας του 90. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία που ήδη έχει περάσει από συνεργασίε, οι διαπραγματεύσει, συγγνώμη, οι διαπραγματεύσει έχουν ολοκληρωθεί και το 97 το Συμβούλιο αποφάσισε να τι παγώσει κάτι που ισχύει ακόμη και σήμερα. Έχουν παγώσει αυτές οι διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 εγγενίασε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Και τότε το Συμβούλιο, εξαιτία των πολιτικών συνθήκων που επικρατούσε στη χώρα, αποφάσισε να μην κρίνει επιλέξιμη τη Λευκορωσία για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Ενώ όλε οι γειτονικέ της χώρε, η Ουκρανία, η Μολδαβία τη Ανατολική Ευρώπη, ανήκουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Πολιτική γειτονία. Εδώ και δύο χρόνια όμως είχαμε κάποιες εξελίξεις στη Λευκορωσία, τις γνωρίζεσαι και το πιο εντυπωσιακό μέτρο που ελήφθη από τον πρόεδρο Λουκασέγκο ήταν η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Και καταρχήν σήμερα δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία. Λέω καταρχήν θεωρητικά, γιατί δυστυχώς ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά το καθεστώς τους είναι συζητήσιμο, αφιλεγόμενο. Παρ' όλα αυτά, το, το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις του καθεστώτος στη Λευκορωσία, αποφυλακίστηκαν πολιτικοί κρατούμενοι, για παράδειγμα, ή υπήρξε κάποια χαλάρωση των περιορισμών προς τους φορείς κοινωνίας των πολιτών, Χάρη σε όλες αυτές τις εξελίξεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε κάποια μέτρα που καταδεικνύουν τη θέλησή της ε, για επανάληψη επαφών με τη Λευκορωσία. Είχαμε καταρχήν κάποιες επισκέψεις του είπα Σολάνα και της ε, Επιτρόπου για τις εξωτερικές ε, σχέσεις της κυρίας Φέραρα Βάλτνερ. Υπήρξαν πολλοί άριθμες ε, επισκέψεις και ανταλλαγές μεταξύ υψηλά ιστάμενων υπαλλήλων και διπλωματών και προσκαλέσαμε τη Λευκορωσία να συμμετέχει στο πολυμερές σκέλος Τη Ανατολική εταιρική σχέση. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό Τσεχική προεδρία το πρώτο εξάμεινο του 2009 και που στόχο έχει την ευάθυνση του πολιτικού διαλόγου με τι χώρες τη Ανατολική Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου και ταυτόχρονα τη σταδιακή του ε, ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκορωσία λοιπόν συμμετέχει στο πολυμερέ τμήμα αυτή τη. Ε, Συμφωνίας Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και μάλιστα συμμετέχει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Συγκεντρώσαμε, συγκεράσαμε τις τέσσερις πλατφόρμες που είναι η η λύθη αυτής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και η Λευκορωσία ήταν πάντα παρούσα και συνέβαλε και συμμετείχε με πολύ θετικό τρόπο. Πριν από λίγες εβδομάδες, οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισαν να παρατείνουν ε, για ένα ακόμη χρόνο τις κυρώσεις ε, προς τη Λευκορωσία, την απαγόρευση κυκλοφορίας για ε, ηθήνοντες και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των ηθινόντων αυτών στις ευρωπαϊκές χώρες και μαζί με την παράταση της, των κυρώσεων ε, αποφάσισαν να παρατείνουν για ένα έτος και την αναστολή των κυρώσεων. Δηλαδή το επόμενο μήνο δεν θα εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση των κυρώσεων γιατί ανεστάλλει για ένα χρόνο αυτό το, αυτή η παράταση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων ζήτησε ταυτόχρονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιήσει δύο τίνα. Καταρχήν να υποβάλει συστάσεις ως προς την πιθανότητα έναρξης διαπραγματεύσεων με τη Λευκορωσία για τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων, βραχυπρόθεσμο θεωρήσεων, έξι ε, ημερών ή βραχυπρόθεσμο. Δηλαδή αυτό που λέμε στα αγγλικά visa facilitation, κάποιες διευκολύνσεις στις θεωρήσεις, στην έκδοση των θεωρήσεων. Επίσης ε, προτάθηκε ένα σχέδιο δράσης, σκιώδες σχέδιο δράσης, δηλαδή να εμπνευστούμε από τα αντίστοιχα σχέδια δράσης με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της, ε, του Νοτιού Καυκάσου στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας και να προσθέσουμε κάτι αντίστοιχο, να προτείνουμε κάτι αντίστοιχο ε, πιο light όμως προς τη Λευκορωσία. Εκεί θα προτείναμε κάποιους στόχους δημοκρατικής μεταρρύθμισης ε, και οικονομικής προσαρμογής και ως αντάλλαγμα της υλοποίησης αυτών των μεταρρυθμίσεων θα προσφέραμε στη Λευκορωσία διάφορα ενδιαφέροντα αντίβαρα. Έχουμε λοιπόν αφενός τη διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων και το Shadow Action Plan. Ένα light σχέδιο δράση για τη Λευκορωσία. Και αν του επόμενου μήνε το καθεστώ του Λουκασέγκο διατρανώσει τη βούλησή του για σταδιακό εκδημοκρατισμό του καθεστώτο και τη κοινωνία, θα κάνει μια χειρονομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση για περισσότερη δέσμευση και σύσφυξη των σχέσεων με τη χώρα αυτή. Πάντως επισημάναμε στις αρμόδιες αρχές της χώρας ότι περιμένουμε τις εξελίξεις σε πέντε κυρίω σημεία. Το πρώτο είναι η απελευθέρωση του πλαισίου λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η διευκόλυνση της ε, μετάδοσης, ειδικά των ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωση στη Λευκορωσία. Επίσης, ε, η αποφυγή σύλληψης πολιτικών κρατουμένων. Τρίτη προϋπόθεση, βελτίωση του συστήματος ε, καταχώρησης ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τέταρτον, τροποποίηση του εκλογικού νόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του ΟΑΣΕ, της ΟΑΣΕ και του ΟΝΤΙΡ. Και πέμπτη προϋπόθεση, η βελτίωση σε ό,τι αφορά το σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης, ώστε να μπορεί η αντιπολίτευση να εκφέρει ελεύθερα τη γνώμη της χωρίς να φοβάται καταστολή καταπίεση. Αυτά προτείναμε λοιπόν στις λευκορωσικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αίσθηση, και αυτή είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την αίσθηση ότι καλό θα ήταν να προχωρήσει η υπογραφή και κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Γιατί η σύναψη μιας συμφωνίας με χώρα εταίρο, ακόμη και αν είναι δύσκολος πελάτης αυτός ο εταίρος, δεν είναι ότι ε, παίζουμε το παιχνίδι του καθεστώτος. Αντίθετα, εφοδιαζόμαστε με ένα μηχανισμό που μας επιτρέπει συνομιλίες και συζήτηση με τη χώρα αυτή για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ακόμη και για τα πιο ακαθόδη και φλέγοντα. Αν έχουμε λοιπόν μια συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασίας με τη Λευκορωσία, θα έχουμε τακτικές ε, συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών, εμπειρογνωμόνων, ή υψηλόβαθμων υπαλλήλων και έτσι θα συζητήσουμε και θα προχωρήσουμε σε θέματα για τα οποία δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτά είναι εν ολίγης ε, τα βασικά σημεία που συνοψίζουν την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Bene, grazie Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίασή σας. Ε, ήδη κάποιοι ζητούν τον λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Παλέξη, Παλέκης. Thank you very much. Ačiū labai. E, buvo tikrai labai įdomu išgirsti. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Ενδιαφέρον. Ήταν ενδιαφέρουσα ήταν ε, η παρουσίαση του αναπληρωτή γενικού διευθυντή και δεν ξέρω εδώ πέρα αν είναι σωστές οι επιλογές ε, οι οποίες έχουν γίνει καθώς η Λευκορωσία ε, με βάση τις δραστηριότητες του Προέδρου της ε, έχει απομονωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση την όθησε προς τα εκεί. Και νομίζω πως οι αλλαγές στη Λευκορωσία είναι μόνο δυνατόν να συμβούν όταν θα έχουμε ευκαιρίες για επαφές σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο στα υψηλότερα, αλλά στο επίπεδο το ανθρώπινο, στο επίπεδο των πολιτισμικών σχέσεων και η ιστορία του 20ου αιώνα μας δείχνει πως ε, η ανατολική πολιτική γειτονία του δυτικού κόσμου μας ε, οδήγησε σε πολλές αλλαγές ε, σε αυτό το τομέα και εγώ θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούν το σωστό δρόμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία τόνισε Πολάκης ε, πως όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία στη Λευκορωσία αυτό το οποίο χρειάζεται είναι διάλογος και νομίζω πως συνεισφέραμε σε αυτό. Η Λιθουανία, η Λετωνία, η Πολωνία, οι γείτονες δηλαδή της Λευκορωσίας υποστηρίζουν και αυτές αυτή την πολιτική. Οπότε θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Ίσως να μην έχετε αρκετό χρόνο να αξιολογήσετε τον νόμο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας ε, για τις αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία. Υπήρξαν επίσημες δηλώσεις που μιλούσαν για τεράστιο βήμα και εγώ θα ήθελα από εσάς να ακούσω την δική σας ανάλυση αυτού του θετικού βήματος των αρχών της Λευκορωσίας. Σωστά αναφέρατε πως οι καλύτερες συνθήκες για τη λειτουργία των ΜΚΟ και της αντιπολίτευσης είναι προαπαιτούμενο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το πώς εκτιμάτε τις ε, επαφές ε, με την αντιπολίτευση, όχι μόνο στο επίσημο επίπεδο, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ δραστήριο εδώ πέρα. Την περασμένη εβδομάδα ο Αλεξάνδρ Μιλινκέβιτς και άλλοι από την αντιπολίτευση ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω και η κυρία Φέρεο Βάλνερ και ο κύριος Σολάν συναντούν ε, ηγέτες της αντιπολίτευσης. Ε, πώς βοηθάτε λοιπόν την αντιπολίτευση, το μεγαλύτερο κομμάτι της αντιπολίτευσης είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ του να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Λευκορωσία και άνθρωποι όπως ο Ανατόλη Λεμπέτσκα και άλλοι ακτιβιστές θεωρούν πως οι επαφές με τις επίσημες αρχές της Λευκορωσίας και η νέα αυτή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύουν το καθεστώς Λουκασάνκο. Αυτές τις ερωτήσεις είχα και σας ευχαριστώ και πάλι για τις πληροφορίες που μας δώσατε. La parola al Προτασίεβιτς, που είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρώπης, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Λευκορωσίας. Είμαι εδώ και δύο χρόνια πρόεδρος αντιπροσωπείας με τη Λευκορωσία, γι' αυτό γνωρίζω αρκετά την ε, κατάσταση και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας. Θα ήθελα να σα πω ότι αν ξεκινήσω από μια ριζοσπαστική έτσι και στεναρή θέση, πριν από ένα χρόνο δέχτηκα μια αλλαγή στην πολιτική απέναντι στη Λευκορωσία. Αντί να κρατήσουμε τη χώρα σε απομόνωση, δέχτηκα να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και επίσημες επαφές, να ενθαρρύνουμε τις αρχές επίσης να σημειώσουν πρόοδο ε, στον δρόμο για τη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, ε, κρίνοντας την κατάσταση μετά από ένα χρόνο, ένα, μισή χρόνο, οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι απογοητευμένος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Καταρχάς, σε σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος Μιγκαρέλη, στον εισαγωγικό του λόγο, καταρχάς η ελευθεροτυπία είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με τη Διεθνή Ομοσπονδία των Δημοσιογράφων και μια έκθεση που έγραψαν πριν από ένα μήνα δεν υπάρχει ακόμα πραγματική ελευθερία για τα πολιτικά κόμματα και για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να λειτουργήσουν ελεύθερα. Κοιτάξτε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στη Λευκορωσία. Την κατάστασή του. Ε, του αρνήθηκαν την επίσημη καταχώρησή του. Και πρόσφατα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήθελε απλώς να αλλάξει όνομα. Ε, αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες με, απέναντι στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, το οποίο του αρνήθηκε την αλλαγή του ονόματο. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Εν συνεχεία, ο εκλογικό νόμο. Πριν από μερικέ εβδομάδε, φαινόταν ε, μια καλή περίπτωση για αλλαγέ. Με βάση την εκπρόσωπο του OECD, της ΩΣΑ, υπάρχει μια τροπολογία του νόμου αυτού που περνάει από την ε, Βουλή της Λευκορωσίας για να εξεταστεί. Αλλά όμως το γραφείο της ΩΣΑ δεν γνωρίζει ποιες είναι αυτές ε, οι αλλαγές. Η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής ε, Επιτροπής στη Λευκορωσία ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο αυτό λαμβάνει υπόψη το 95% των συστάσεων που πρότεινε η ΟΝΤΙΡ και η ΟΑΣΕ αλλά δεν ξέρουμε αν είναι πιο σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές. Και παρά μια γραπτή συμφωνία μεταξύ της Κεντρικής εκλογική επιτροπή και του γραφείου τη ΟΝΤΙΡ το περασμένο Φεβρουάριο, ότι πριν περάσει αυτό το νομοσχέδιο από τη Βουλή θα γίνει συζήτηση ξανά με το γραφείο τη ΟΝΤΙΡ, δεν έγιναν καθόλου διαβουλεύσεις για τι τις αλλαγές αυτές. Επομένως, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα της αλλαγής του εκλογικού νομού. Και τέλος, όπως είπε ο κύριος Μιγκαρέλη, υπάρχουν 10 άτομα ακόμα, τα οποία θεωρούνται από τη Διεθνή Αμνηστία ως φυλακισμένοι συνείδηση στη Λευκορωσία. Ο ένας από αυτούς, μάλιστα, είναι ακόμα φυλακισμένος, ο κύριος Ντόψκι. Θα ήθελα να αναφέρω το όνομά του, παρακαλώ. Τέτοια θέματα λοιπόν τίθενται. Τέτοια θέματα υπάρχουν. Ε, σε αυτή τη νέα λοιπόν στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και ο διάλογος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ο οποίος έχει ξεκινήσει. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου. Υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. Και δεύτερον, πριν από λίγο, πριν από λίγες μέρες, όταν είχα μια ανταλλαγή απόψεων με το νέο, είπα το εκπρόσωπο για τις εξωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ε, Βαρόνη Άστον, μίλησε για μια ήσυχη διπλωματία. Με ανησυχεί όμως ότι αυτή η ήσυχη διπλωματία στην περίπτωση της Λευκορωσίας μπορεί να οδηγήσει σε σιωπή για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις αυτών. Ε, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, όχι μόνο για μας, αλλά κυρίως για την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας υπό την αιγίδα του κυρίου Μιλίνκεβιτς που υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, μπορεί να χάσουν έτσι την αξιοπιστία τους στην ε, κοινωνία της Λευκορωσίας. Μια και η πολιτική αυτή δεν θα δημιουργήσει πραγματική αλλαγή στην κοινωνία. Αλλά και δεύτερο, πολύ πιο σημαντικό, μπορεί εκείνος να χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμά αν ε, οι δικές μας πολιτικές απλώς παρακάμπτουν τα, την αντιπολίτευση και δεν τη συμπεριλαμβάνουν σε αυτό το διάλογο. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι Δευτέρα ο κύριος Μπερλουσκόνη επισκέφθηκε επίσημα το Μίνσκ. Είναι η πρώτη φορά που ένας Ευρωπαίος ηγέτης πήγε στο Μίνσκ. Πολύ ωραία, μια χαρά. Αλλά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του δεν συνάντησε την ε, δημοκρατική αντιπολίτευση. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι κύριε Μιγκαρέλη εσείς δεν το υποστηρίζετε αυτό και ότι στο μέλλον θα αποφευθεί κάτι τέτοιο. Δεν θα το ξαναεπαναλάβει άλλος Ευρωπαίος ηγέτης. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Μετά από αυτές τις δύο παρεμβάσεις έχουμε τους επόμενους που ζητούν το λόγο. Και συνεχεία μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη Συρία και το Αφγανιστάν. Ακριβώ γι' αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλοί ομιλητέ, θα ήθελα ο καθένα να περιοριστεί σε δύο λεπτά. Ο πρώτο που θα ακολουθήσει τώρα είναι ο κ. Σούλτσα. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Μιλήσατε για τις πιθανότητες που εξερευνούνται πάρα πολύ εντατικά περί μιας συμφωνία γειτονίας. Η μία εταιρική σχέση εμποδίζει την άλλη. Πώς αξιολογείτε την Τελωνιακή Ένωση Ρωσίας-Λευκορωσίας. Και ενώ διαπραγματευόμαστε εταιρική σχέση με την Ρωσία και το ζήτημα που τίθεται είναι η ένταξη στον ΠΟΕ της Ρωσίας

Θα ήθελα να υποστηρίξω τα λόγια του κυρίου Προτασέβιτς ότι ήρθε η στιγμή να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με την αντιπολίτευση. Γιατί αν παρακάμψουμε την αντιπολίτευση στις πολιτικές σχέσεις με τη Λευκορωσία, έχει επίγνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι αποτελέσματα θα έχει. Πιστεύετε ότι θα οδηγήσει κάτι τέτοιο στην ενίσχυση του Λουκασέγκο ή στην ανατροπή του θα πρέπει να μην δώσουμε δίκαιο στο καθεστώ του Λουκασέγκο. Θα πρέπει να υπάρξει σαφή και απερίφραστη δήλωση και του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είστε πεπισμένοι ότι αυτή η κατάσταση σχέσεων με την αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα, δηλαδή οι πολιτικέ σχέσει που έχουμε με την αντιπολίτευση σήμερα, είναι αρκετέ και ενισχύει το κύρο. Γιατί θέλουμε ακριβείς πληροφορίες. Τι μορφή έχουν οι ευρωπαϊκές σχέσεις με την λευκορωσική αντιπολίτευση. Όταν ο κύριος Σολάνα και η κυρία Φεραίρο Βάλτνερ επισκέφθηκαν ε, τη Λευκορωσία, συναντήθηκαν με μέλη της αντιπολίτευσης. Γιατί σίγουρα το πήγε ο Μπερλουσκόνη, δεν συναντήθηκε με μέλη της αντιπολίτευσης. Όταν έχετε ε, με τις λευκορωσικέ αρχές, θα πρέπει ταυτόχρονα να συναντάτε και μέλη της αντιπολίτευση. Και αν δεν μου απαντήσετε συγκεκριμένα θα σα θέσω και γραπτή λεπτομερή απάντηση, γιατί νομίζω ότι έτσι θα κριθεί το κύρος της αντιπολίτευσης. Η, Ευρωπαϊ... η λευκορωσική αντιπολίτευση θέλει ε, αποδείξεις, ε, θέλει χειρονομίες για να δείξει ότι είναι έγκυρη αντιπολίτευση, ότι έχει κάποια έγκλη και κύρος. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα κρυθεί από τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ενδιαφέρει πολύ η εκτίμηση που κάνει για τα πράγματα αυτά ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα του εκλογικού νόμου έχω την εντύπωση και θα ήθελα παρακαλώ να είναι μονολεκτικό το σχόλιο σας. Δεν έχει νόημα να επενούμε το Λουκασέγκο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Το θέμα είναι να γίνουν πραγματικά ελεύθερες εκλογές, γιατί η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου δεν σημαίνει αυτόματα και διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών. Μερικές φορές είναι ένα παραπέτασμα που ε, θεσπίζεται για τη δημιουργία εντυπώσεων και παρόλα αυτά θέλει να διοργανώσει μη ελεύθερες εκλογές. Ε, με τι κριτήρια λοιπόν αξιολογούμε έναν εκλογικό νόμο. Θα ήθελα την ε, γνώμη του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρικέν έχει το λόγο. Παρακαλώ, συνοπτικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο ρόλος να λογοκρίνω τους ομιλητές. Αλλά είναι θέμα δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε θερμά κύριε Μιγκαρέλη για τη γενική επισκόπηση που μας κάνατε της κατάστασης της Λευκορωσίας. Εγώ έχω μία ερώτηση για την οικονομική κατάσταση της Λευκορωσίας. Ποιε είναι οι πληροφορίες και οι γνώσεις σα για την κατάσταση της λευκορωσικής οικονομίας, ειδικά στο πλαίσιο τη παγκόσμια χρηματοπιστωτικής κρίση. Δεύτερον, οι λευκορωσικές αρχέ. Ε, από ό,τι φαίνεται έκανα κάποια βήματα για την απελευθέρωση της οικονομίας τα τελευταία χρόνια και μάλιστα ισχυρίζονται ότι έχουν εξασφαλίσει μεγαλύτερη ελευθερία στο αλλοδαπό κεφάλαιο. Ε, είναι λυθείς αυτές οι δηλώσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία του αλλοδαπού και μεγαλύτερη διείσδυση ευρωπαϊκών εταιριών στη λευκορωσική οικονομία. Πρόσφατα έγινε μια κοινή δήλωση από Ρωσία, Λευκορωσία και Καζακστάν ότι τρεις χώρες ως Τελωνιακή Ένωση από κοινού θα προσχωρήσουν στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Τι είναι αυτό, προπαγάνδα ή υπάρχει κάτι σοβαρό και συγκεκριμένο πίσω από αυτή την κοινή δήλωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Βιγγένιν. Ευχαριστώ είμαι πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου στην συνέλευση της Euronest που δεν έχει ακόμη ε, ξεκινήσει λειτουργίες, αλλά είμαστε σε φάση ετοιμασία. Και ένα βασικό θέμα που έχουμε είναι η συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτή τη συνέλευση. Το Κοινοβούλιο δεν είναι έτοιμο να αναγνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας έχει εκλεγεί, καλώντας τα μέλη του Κοινοβουλίου της Λευκορωσίας να συμμετάσχουν πλήρως στη Euronest. Έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις ήδη φέτος. Θα αναθεωρήσουμε αυτές τις αποφάσεις και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποια μικρά βήματα, αλλά μέχρι να εκλεγεί δημοκρατικά το Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να, συμμετάσχουμε, να συμμετάσχουν οι βουλευτές της Λευκορωσίας σε ίση βάση στην Euronest. Τώρα, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά έχω μία ερώτηση. Ε, πόσο αξιολογείται τη συμμετοχή τη Λευκορωσία στην εταιρική σχέση προ Ανατολά και κατά την άποψή σα, ε, ποια είναι η δέσμευση που έχω αναλάβει για να παραμείνουν τμήμα αυτή τη πολιτική. Αυτή η μη πρόσκληση προς τη Λευκορωσία θα μπορούσε να θέσει ε, αμφιβόλο την όλη διαδικασία, γιατί φυσικά υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των ανατολικών χωρών. Και πιστεύετε ότι είναι σόφρον από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθήσει να αναπτύξει μια πιο συντονισμένη πολιτική μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν απέναντι στην Λευκορωσία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ορισμένες πτυχές αυτής της πολιτικής, που έχει ήδη μπει στα σκαριά. Το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτή την πολιτική, αλλά φυσικά παράλληλα υπάρχουν ε, κάποια θέματα αρχών, τα οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας από τη μία, από την άλλη και εσείς όμως πιστεύω ότι χρειάζεται και τη δική μας ε, υποστήριξη για να τελεσφορήσει αυτή η εταιρική σχέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Το 2002 ε, για πρώτη φορά μπήκα στην Επιτροπή Λευκορωσίας και Μολδαβίας και Ουκρανίας. Ε, θυμάμαι ότι τότε γνώρισα τον κύριο Μιγκαρέλη και είναι πραγματικά πεπειραμένος παρατηρητής στα θέματα της ε, Λευκορωσίας. Πιστεύω ότι η πολιτική απομόνωση που προωθούν τα κράτη-μέλη και οι Ηνωμένε Πολιτείε στην πραγματικότητα την απομονώνει, ε, δεν δίνει αποτελέσματα ε, και νομίζω ότι το καρότο και το μπαστούν είναι μια καλύτερη προσέγγιση. Ο κύριος Λουκασέγκο ε, είναι πονηρή αλεπού. Έχει περάσει από τη Σοβιετική εποχή, δεν είναι δημοκράτης και ποτέ δεν θα γίνει, αλλά σίγουρα καταλαβαίνει από πολιτική και επομένως θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη σοβαρά. Πρώτη ερώτηση. Ε, προέκυψε στο ε, ε, Είναι η, τα στρατιωτικά γυμνάσια της Λευκορωσίας με την Ρωσία, όπου δεν υπήρχαν καθόλου παρατηρητές από τον ΝΑΤΟ. Αυτό μου φαίνεται προκλητικό. Και το σενάριο που σκιαγραφήθηκε ήταν ε, εισβολή από Λιθουανούς ε, τρομοκράτες. Αυτό είναι πραγματικότητα, η φαντασία δεν ξέρω. Αυτό άκουσα πάντως. Εν περιπτώσει, πώς το σχολιάζετε αυτό, αυτά τα σενάρια, αυτά τα γυμνάσια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό που συζητούμε σήμερα είναι πολύ πιο σημαντικό στα πλαίσια της τελευταίας επίσκεψης ε, των ε, της αντιπροσωπείας της αντιπολίτευσης με επικεφαλή τον κύριο Μιλινκέβιτς και πολλούς άλλους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Και εκεί μας επισήμαναν όχι μόνο την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση της αντιπολίτευσης στην Λευκορωσία, αλλά και το θέμα της ελευθεροτυπίας, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, αλλά και Μία λιδία λίθος ε, για το τι συμβαίνει στην Λευκορωσία είναι οι μελλοντικέ ε, περιφερειακές και δημοτικές ε, εκλογές. Γιατί θα φανεί εκεί αν ο εκλογικός νόμος που είναι θεωρητικά καλός θα εφαρμοστεί και εμπράκτος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά πόσο όντως η αντιπολίτευση θα συμμετέχει και θα φανεί και στα αποτελέσματα των εκλογών. Η οικονομική κατάσταση της Λευκορωσίας σίγουρα δεν είναι εύκολη και αυτή η οικονομική κατάσταση φυσικά σχετίζεται με, την, με τις αστρονομικές τιμές των πρώτων υλών και του φυσικού αερίου μεταξύ άλλων που είναι υψηλές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε το θέμα δεν είναι να βοηθήσουμε μόνο σε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να βοηθήσουμε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Γιατί αυτή είναι η γνώμη των μελών τη αντιπολίτευση. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο να δοθεί αρρωγή, αλλά να συνδυαστεί αυτή με κάποιες θετικές εξελίξεις στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών της αντιπολίτευσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση. Και τελευταία φράση. Το θέμα της μείωσης του κόστους ε, των θεωρήσεων για τους ελευκορώσους πολίτες. Ο Επίτροπος Μπαρό είπε ότι σήμερα με βάση τις συμφωνίες δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των τιμών των θεωρήσεων. Πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρόλα αυτά μπορεί να σημειωθεί κάποια πρόοδος εκεί. κολέγα ονορεύλε Ο κ. Παντσέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας ε, κύριε Μιγκαρέλη. Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε μια χώρα όπως η Λευκορωσία να μπει στο δρόμο της, του εκδημοκρατισμού και της, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι και τα ερωτήματα που σας θέτουμε, ακριβώς γι' αυτό τα θέτουμε. Ε, επίσης, και αυτός ο εφημισμός που ονομάζεται εκλογικός νόμος, στην πραγματικότητα εκφράζει την κατάσταση της δημοκρατίας αυτή ε, τη χώρα. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Και θα ήθελα να καταλάβω, υπενθυμίζοντας λίγο αυτό που είπε ο κύριος Ποτατσίεβιτς, πώς εκτιμάται από πλευράς Κομισιόν την ε, πρόσφατη επίσκεψη του Ιταλού Πρωθυπουργού με την συνάντηση που είχε με τον Λουκασέγκο, που τον οδήγησε τον Λουκασέγκο να πει στον τύπο ότι υπάρχει ένα άνοιγμα της Ευρώπης απέναντι στη Λευκορωσία. Τώρα, προσοχή, όχι παρεξηγήσεις. Φυσικά, η κάθε χώρα έχει το προνόμιο να κανονίζει τις επισκέψεις της στο εξωτερικό. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπήρξε κάποια διαβούλευση μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν και αν ε, δόθηκε εντολή <laughs> ενδεχομένω στον κύριο Μπελουσκόνη να διανοίξει νέες διπλωματικές οδούς και αν όχι, αν δεν συνέβη κάτι τέτοιο, πώς κρίνει η Κομισιόν αυτή την εκτίμηση, αυτή την επίσκεψη. Προκειμένου να μην έχουμε μια εξωτερική πολιτική όπου καθένα κάνει ό,τι θέλει. Κάτι άλλο. Καλό θα ήταν σήμερα το πρωί να χαρωτήσει την Βαρόνη Άστον για της χαρωτήσει αυτό το, αυτό το θέμα. Ε, δεν μπόρεσα να θέσω αυτό το ερώτημα στην κυρία Άστον. Ε, το θέτω σε εσά. Ευχαριστώ, κύριος Μίνσκι. Εγώ έχω πάει πολλές φορές στην Λευκορωσία και γνωρίζω την κατάσταση στη χώρα. Σήμερα όλοι μπορούν να πούν πως ε, εγώ εκπροσωπώ, ο καθένας δηλαδή, εκπροσωπεί την αντιπολίτευση στην ε, Λευκορωσία. Και ε, ο κύριος Μιλικέβιτς τώρα 300 άτομα εκπροσωπεί. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Η πλειοψηφία δεν υποστηρίζει την αντιπολίτευση. Οπότε έχω μία ερώτηση. η Κομισιόν και το Συμβούλιο σκοπεύουν να εντείνουν τις επαφές με την κυβέρνηση της χώρας. Η τελευταία παρέμβαση, ε, ο κύριος Σαρλάκη. Ε, παρετήστε, άρα το λόγο έχει ο κύριος Μιγκαρέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις και για όλα τα σχόλια. Ε, θα απαντήσω σε κάθε ερώτηση ε, εντάχει η νέα εκλογική νομοθεσία καταρχάς. Δεν είμαστε σε θέση προς το παρόν να σας πούμε ποια είναι τα αποτελέσματα του δικού μας προβληματισμού, γιατί αυτή η νέα νομοθεσία υπάρχει εδώ και λίγες μέρες μόλις. Αλλά οι παρατηρητές οι οποίοι κοίταξαν το νέο νόμο εκ του σύνεγγης ε, λένε ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι δική μας αξιολόγηση, το επαναλαμβάνω, γιατί δεν είμαστε ακόμη σε θέση να σας την ανακοινώσουμε. Αλλά διάφοροι παρατηρητές ε, εξέτασαν αυτό το νέο νόμο και λένε ότι μάλλον συνιστά έναν εκδημοκρατισμό και δημιουργεί κάποιες πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις στην ομαλή διεξαγωγή των ε, εκλογών. Ο κύριος Κόβαλ λέει ότι καλό είναι να υπάρχει ένας νέος εκλογικός νόμος, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Προφανώς. Δεν αρκεί ύπαρξη του νέου νόμου. Είναι ένα πρώτο βήμα μόνο. Καταρχάς ζητάμε από αυτή τη χώρα να περάσει ένα νέο νόμο ε, με βάση τις συστάσεις του, της ΟΝΤΙΡ και του, της ΟΑΣΕ και συνεχεία να την εφαρμόσει αυτή η χώρα. Και αν δεν την εφαρμόσει στις ε, ε, δημοτικές εκλογές που θα γίνουν την Άνοιξη του 2010, προφανώς θα πάρουμε κι εμείς ε, ένα μήνυμα. Αλλά τα πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα είναι ένα βήμα σωστή κατεύθυνση. Δεν αρκεί, αλλά πρέπει να το σημειώσουμε και να το καταγράψουμε ως τέτοιο. Ως τέτοιο. Επαφές με την αντιπολίτευση. Ανασκευάζω τα όσα είπε κάποιος βουλευτής, δηλαδή ότι αγνοούμε την ε, αντιπολίτευση και ότι δεν ερχόμαστε σε επαφή. Είναι λάθος. Σε κάθε επίσκεψη που γίνεται από τη Γραμματεία του Συμβουλίου και υπαλλήλου Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντούμε κάθε φορά τα μέλη της ε, αντιπολίτευσης. Και όταν ο κ. Σολάνα πήγε και όταν η Επίτροπος Φέρο Βάλτνερ επίσης πήγε, έκανε το ίδιο. Είναι λάθος λοιπόν αυτό που λέγεται. Κάθε φορά συναντούμε την αντιπολίτευση σε κάθε επίσκεψη. Επίσης εδώ και χρόνια, ε, από το 97 χρηματοδοτούμε τους ανεξάρτητους φορείς των ΜΜΕ, των κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των διαφόρων συνδικάτων και ενώσεων. Μας κατηγορείτε ότι δεν χρηματοδοτούμε πολιτικά κόμματα, αλλά εξηγήσαμε ότι λαμβάνοντας υπόψη το χρηματοδοτικό κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε ε, πολιτικά κόμματα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αλλά υπάρχουν ε, διάφορα πολιτικά ιδρύματα των κρατών μελών που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω ότι δεν αγνοούμε την αντιπολίτευση. Οι υπάλληλοι μας συναντώνται συστηματικά με μέλη της αντιπολίτευσης. Και την επόμενη φορά που ε, ο κύριος Μιλίνκεβιτς ε, ε, θα είναι παρόν και θα συναντηθείτε, ρωτήστε τον. Η αντιπολίτευση σε μεγάλο βαθμό χρειάζεται μια ενεργητική πολιτική. Προσοχή λέω, σε μεγάλο βαθμό. Μας λέει, εντάξει, ελάτε, ξεκινήστε προγράμματα ε, συνεργασίας, στείλτε εμπειρογνώμονες. Για αυτούς είναι σημαντικό να μην είναι απομονωμένοι. Είναι σημαντικό να είναι σε επαφή με τον έξω κόσμο. Αυτό μας το λέει η μεγάλη πλειοψηφία της αντιπολίτευσης. Φυσικά μας λέει, ε, μην είστε και κορόιδα, ε, δείτε ποιες είναι οι νέες, τα τελευταία τεχνάσματα του Λουκασέγκο. Δείχνει αυτή την καλή θέληση γιατί, γιατί στριμώχνεται τρομερά για οικονομικούς λόγους και όχι γιατί ξαφνικά έγινε δημοκράτης. Αλλά μας λένε, εποφεληθείτε από αυτό το άνοιγμα, ελάτε, μην μας αφήνετε στριμωγμένου στον τοίχο και εξασφαλίστε την επίσκεψη πολλών Ευρωπαίων πολιτών στη Λευκορωσία για να έχουμε και εμείς επαφές. Η αντιπολίτευση πρέπει να πούμε ότι είναι διαιρεμένη. Αυτό συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό ε, στη μεγάλες εκλογικές του Λουκασέγκο. Δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι υπάρχει εκλογική νοθεία. Υπάρχουν δύο στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το πρώτο είναι ότι η αντιπολίτευση είναι διαιρεμένη και το δεύτερο και ορισμένοι το είπαν, ε, θα αναπηδήσουν μάλλον, ε, ότι μέχρι στιγμή το μέσο επίπεδο ζωή του μέσου κατοίκου ήταν ανώτερο από το μέσο βιωτικό επίπεδο γειτονικών χωρών. Είναι δεδομένο, δεν το λέω εγώ. Το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο. Και αυτό σε κάποιο βαθμό εξηγεί το γεγονός ότι ακόμη και αν υπήρχαν δίκαιες εκλογές και μεινοθευμένες, τα αποτελέσματα δεν θα ήταν άρδιν διαφορετικά. Ο κύριος Ποτάσιεβιτς μας ρωτάει να, μας πει ποια είναι να του πούμε ποια είναι η αξιολόγηση για αυτό το άνοιγμα, από αυτό το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δύο χρόνια. Έχετε δίκιο, δεν υπάρχουν θεαματικές αλλαγές. Έχουμε πει και ξαναπεί ότι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες ξεκίνησαν δεν είναι ούτε ε, συστηματικές, ούτε ε, μονοσήμαντες. Και όπως είπε ο Τάνοκ, όμως ε, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η εναλλακτική λύση είναι η απομόνωση της χώρας. Η απομόνωση δεν οδηγεί πουθενά. Παρότι θεωρούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι δειλές, ε, ανεπαρκείς, νομίζουμε ότι θα πρέπει να τις ενθαρρύνουμε εφαρμόζοντας αυτή την πολιτική του ε, μπαστούνιου και του καρότου. Μας λέτε ότι δεν υπάρχει ελευθερία για την αντιπολίτευση. Έχετε δίκιο, το επιβεβαιώνω. Είναι επικίνδυνο να είναι κανείς αντιφρονών. Είναι δύσκολο ε, μια ανεξάρτητη εφημερίδα να πουλιέται ανοιχτά και είναι δύσκολο για μια μη κυβερνητική οργάνωση να καταχωρηθεί ως τέτοια. Ε, είναι αλήθεια, αλλά έγιναν κάποια δειλά βήματα προς σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε. Θα τελεσφορήσουν, δεν το ξέρω. Πρέπει να πάρουμε ένα ρίσκο. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο επικίνδυνο να καθίσουμε άπραγοι και να τους κατακεραυνώσουμε παρά να βοηθήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, για τα οικονομικά θέματα. Άνοιξε κάπως το καθεστώς, έδειξε άνοιγμα, γιατί για πρώτη φορά εδώ και 12-13 χρόνια υπάρχουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η τιμή του ρωσικού αερίου αυξάνει κάθε τόσο, τακτικά, και επομένω υπάρχει πρόβλημα. Γιατί φυσικά αυτή η οικονομία ε, επιδοτείται από τις τεχνητέ τιμέ ε, του αερίου που χορηγούσε η Ρωσία. Και επίσης υπάρχει και το, και το πρόβλημα που υφίστανται λόγω της παγκόσμιας κρίσης. Επομένως, ε, αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν ε, διαπραγματεύσει με το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο για τη βοήθεια του και ζητάνε και μακροοικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν πρότεινε στο Κοινοβούλιο να δώσει τέτοια οικονομική βοήθεια 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, συζητιέται βέβαια αυτό το θέμα, δεν είναι δεδομένο και θα το συνδυάσουμε με αυστηρές προϋποθέσεις, με βάση αυτά που πριτανεύει και το Διεθνές Αμεσματικό Ταμείο. Κάθε φορά αυτό γίνεται. Η κατάσταση η οικονομική και μακροοικονομική είναι πολύ δύσκολη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα και προφανώς γι' αυτό υπάρχει και ένα άνοιγμα των ηθινών του καθεστώτος. Μας ρωτάτε αν η Τελωνιακή Ένωση που προσπαθεί να δημιουργήσει η Λευκορωσία με τη Ρωσία και το Καζακστάν μπορεί να έχουν επίπτωση στη σχέση μας με τη χώρα αυτή. Εδώ και χρόνια υπάρχει μια τελωνιακή ένωση μεταξύ της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Αλλά δεν λειτουργεί. Δεν δίνει αποτελέσματα. Είναι όπως όλες οι συμφωνίες που υπογράφτηκαν στα πλαίσια της ε, ΚΑΚΑ. Υπογράφηκαν πάρα πολλές ε, συμφωνίες, αλλά στην πράξη λίγα έχουν γίνει. Είναι μια τελωνιακή ένωση που έχει μείνει κενό κενή περιεχομένου. Ε, οι Ρώσοι όταν ε, εισάγουν προϊόντα από τη Λευκορωσία ακόμα βάζουν τελωνιακούς δασμούς. Αύριο μεθαύριο, όταν θα υπάρχει αυτή η τελωνιακή ένωση με το Καζακστάν, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα έχει επιπτώσει σε εμά. Δεν θα μα εμποδίσει να υπογράψουμε τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία και θα μα εμποδίσει να προχωρήσουμε αυτό το σχέδιο δράση στην ε, πολιτική αυτή γειτονία. Το πρόβλημα είναι όταν έχουν αυτή τελωνιακή ένωση και θέλουν να έχουν μαζί μα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη φάση διαπραγματεύση ε, τέτοια συμφωνία με τη Λευκορωσία. Το πρόβλημα όμως τίθεται με τη Ρωσία, το ξέρετε κυρία μου. Γιατί η Ρωσία αποφάσισε τώρα να ενταχθεί στο, α, στον ΠΟΕ στα πλαίσια της Τελωνιακής Ένωσης με το Καζακστάν και την α, Λευκορωσία. Ε, εκεί έχουμε πρόβλημα. Ε, θα είμαι πιο σύντομος, ναι. Η συμφωνία, η συμμετοχή μάλλον ε, στην ε, συμφωνία ανατολικής γειτονίας. Έχουμε την ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια, οικονομική ένταξη και επαφή των λαών. Ε, κάθε φορά ήρθαν σε επίπεδο υπουργικό με πολλούς εμπειρογνώμονες και θέλουν να συμμετάσχουν. Ε, υπάρχει βέβαια ε, κίνδυνος ενό προβλήματος αν αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της Απχασίας και της νότιας αιτίας. Αν αναγνωρίσουμε με τη Ρωσία την ανεξαρτησία αυτών των περιοχών, έχουμε πρόβλημα με τη Γεωργία, που είναι τμήμα της σχέση σχέσης αυτής. Τώρα, για, για τα στρατιωτικά γυμνάσια, κύριε Τάνοκ, με δυσκολεύετε εδώ. Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Ε, στη τελευταία γκάρκ, ο Πολωνός ε, Υπουργός μας ε, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτά τα γυμνάσια στη Λευκορωσία για τους λόγους που αναφέρατε. Τι, τι γνώμη έχω, τι να σας πω. Μακάρι να μην γινόταν αυτά γυμνάσια. Είναι ανησυχητικά φυσικά. Και το γνωστοποιούμε αυτό στην ε, Λευκορωσία. Τώρα, το ερώτημα του κύριου Παντζέρη για την επίσκεψη του Μπερλουσκόνη. Ε, καταλαβαίνετε ότι ένας υπάλληλος της Κομισιόν δεν θα ήθελε να σχολιάσει ε, τα πεπραγμένα των αρχηγών ε, κρατών και κυβερνήσεων. Τώρα, για το ότι θα πρέπει η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συντονίζονται καλύτερα μεταξύ της Κομισιόν και του Συμβουλίου, το πρόβλημα θα ρηθεί σε λίγε εβδομάδες. Τώρα για το Κοινοβούλιο κάθε φορά που το επιθυμείτε θα ερχόμαστε εδώ και θα λογοδοτούμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε και θα λαμβάνουμε υπόψη τι ανησυχίε και τι συστάσει σα για να προσαρμόσουμε αναλόγω τι στρατηγικέ μα. Ευχαριστώ νομίζω ότι κάλυψα ή ελπίζω τουλάχιστον να κάλυψα τι περισσότερε ερωτήσει. Θέλετε κάτι Διαδικαστικό θέλετε, ναι. Υπήρξε μια παρεξήγηση. Φυσικά και γνωρίζω ότι γίνονται επαφέ με την λευκορωσική αντιπολίτευση μεταξύ Σολάνα και Φέρερ Βάλτερ και το εκτιμώ ιδιαίτερω. Είναι δικαστικό το θέμα σα. Μια μου, μια μου. Επειδή με παρανόησε, ακριβώ επειδή με αφήσετε να ολοκληρώσω όταν έθετα την ερώτηση, δεν κατάλαβα να πληρωτήσει Γενικώ Διευθυντή, εγώ ξέρω ότι γίνονται επαφέ. Σα ρώτησα αν τι κρίνετε επαρκή, αν είναι ή μήπω ε, δεν είναι αρκετά έντονε. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Γι' αυτό υπήρξε και παρεξήγηση. Φυσικά πάντα ε, υπάρχει δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Και ποτέ δεν βοηθάμε αρκετά τόσο θαραλέου ανθρώπου ε, που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Πάντα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ για την πρώτη σας παρέμβαση. Θα περάσουμε τώρα στη Συμφωνία ε, Συνεργασίας με τη Συρία. Σύνδεση, συγγνώμη, με τη Συρία. Θα μπορούσα να κάνω μια πρώτη γενική παρουσίαση ως ε, πρόεδρος, αλλά δεν χρειάζεται να την κάνω. για να εξοικονομήσουμε χρόνο θα θα σα δώσω κατευθείαν το λόγο. Θα είμαι πραγματικά επιγραμματικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ξέρετε, διαπραγματεύτηκε μεταξύ 2000 και 2004 μια συμφωνία σύνδεση με τη Συρία. Το 2004 ολοκληρώσαμε τι διαπραγματεύσει, αλλά εξαιτία κάποιων πολιτικών δυσκολιών που υπήρχαν τότε στη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση-Συρία, το Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να μην υπογράψει και να μην κυρώσει αυτή τη συμφωνία σύνδεση με τη Συρία. Το 2008, δηλαδή πέρυσι, και μετά τις εξελίξεις της Συριακής πολιτικής απέναντι στις γειτονικές της χώρες, αποφασίστηκε από το Συμβούλιο ότι ήταν τώρα σκόπιμο να συνεχιστούν οι συζητήσεις με τη Συρία και έγινε μια ενημέρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης στα τέλη του 2008 Πήγαμε στη Δαμασκό το Δεκέμβριο του 2008 για τη μονογραφή της συμφωνίας και το πρώτο εξάμεινο του 2009 μεταφράσαμε τη συμφωνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγξαμε την νομική του ακρίβεια, ώστε να μην δώσει λαβή για προσφυγές και η Συρία υιοθέτησε μια μονομερή δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μονομερή δήλωση για το υπό ποιε προποθέσει θα μπορούσε να ανασταλεί αυτή η συμφωνία λόγω καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Σουηδική Προεδρία κάλεσε τον Νοέμβριο τον Σύριο Υπουργό ε, για να υπογράψει στις Βρυξέλλες τη συμφωνία. Η απάντηση του Υπουργού Μοαχαλέμ ήταν ότι δεν, δεν είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε αμέσως αυτή τη συμφωνία. Θα πρέπει να την εξετάσουμε πιο διεξοδικά, πιο προσεκτικά και εν συνεχεία θα σας πούμε αν θέλουμε να υπογράψουμε την έκθεση αυτούσια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις Συριακές Αρχές να τους βοηθήσουν στην αξιολόγηση της συμφωνίας, αλλά οι Σύριοι μας είπαν ότι προς το παρόν δεν έχουμε ανάγκη. Θα κάνουμε τη δική μας αξιολόγηση και θα υποβάλουμε στον πρόεδρο Ασάντ τα αποτελέσματα της αξιολόγησής μας τον επόμενο Μάρτιο. Και γνωρίζω ότι στο μεταξύ ξεκίνησαν διαβουλεύσεις με γειτονικέ χώρες που ήδη έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Αλγερία, η Ορδανία και η Αίγυπτος. Τώρα, για ποιο λόγο θεωρούν οι Σύροι ότι δεν είναι επίγουσα η υπογραφή της συμφωνίας, πιστεύω ότι τρεις είναι οι Καταρχήν, θέμα πρωτοκόλλου. Δώσαμε δέκα ημέρες στον Σύριο Υπουργό για να έρθει στις Βρυξέλλες. Το έκρινε ως τελεσίγραφο. Δεν θεώρησε ότι είναι ε, αποδεκτή μια τέτοια προϋπόθεση. Μας είπε εδώ, μας αφήνατε να περιμένουμε τέσσερα χρόνια και μας δίνετε δέκα μέρες για να έρθουμε να υπογράψουμε στις Βρυξέλλες. Ε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και κάπου το καταλαβαίνουμε. Δεύτερος λόγος, οι Συριακές αρχές ε, ενοχλήθηκαν από τη μονομερή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόλο που η δέσμευση αυτή δεν δεσμεύεται, η δήλωση αυτή δεν δεσμεύει τη Συρία, θεώρησαν ότι μια τέτοια δήλωση συνιστά δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση της Συρίας απέναντι στις υπόλοιπες χώρες ε, της Μεσογείου, γιατί τέτοιες μονομερείς δηλώσεις δεν έχουν επισυναθεί σε καμία άλλη συμφωνία σύνδεσης. Αλλά υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι. Οι Σύριοι θεωρούν ότι από οικονομική άποψη η συμφωνία αυτή σύνδεση δεν θα τους είναι ιδιαίτερα επωφελής. Βραχυπρόθεσμα μάλιστα θα υπάρξουν κάποια, φορο... κάποια απώλεια φορολογικών εσόδων, ε, θα υποστούν ε, το στιγνό ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις τους σε κάποιους τομείς που ήδη είναι ευάλωτοι. Ίσως υπάρξει αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών ε, προς τη Συρία για ορισμένους τομείς, ενώ το αντίθετο αύξηση των εξαγωγών της Συρίας είναι μάλλον απίθανο βραχυπρόθεσμα. Επίσης μας ζήτησαν ενισχυμένη χρηματοπιστωτική αρρωγή για να βοηθήσουμε τη Συρία να εξυγχρονιστεί κατά την προσπάθεια εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Εμείς εξηγήσαμε στη Συρία ότι μέσω και μακροπρόθεσμα η εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας εφόσον συνδυαστεί με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη Συρία προκειμένου να ανοίξει η οικονομία θα είναι επωφελής για τη χώρα μέσω και μακροπρόθεσμα και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε στη Δαμασκό στην επόμενη συνάντηση να υποστηρίξουμε με επιχειρήματα τη θέση μας ώστε να πείσουμε τους Σύριους να υπογράψουν γιατί για μας είναι σημαντικό να έχουμε μια συμβατική βάση για να ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις μας με τον τόσο σημαντικό εταίρο που είναι η Σύρια. Αυτά είναι ολίγης μια ανακεφαλαίωση της κατάστασης με τη Σύρια. Καλώς. Φυσικά υπάρχει πάλι εκτενής κατάλογος ομιλητών. Πρώτα θα το λόγο στον εισηγητή για τη Συμφωνία Σύνδεσης και ταυτόχρονα αντιπρόεδρο Μποντί. Euh, Κύριε Μικαρέλη, χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που συζητούμε για αυτή την ε, Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Συρίας. Γιατί είχαμε και άλλες συμφωνίες σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Αραβικών χωρών, είτε νοτίως της Μεσογείου, είτε ανατολικά. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της συμφωνίας σύνδεσης με τη Συρία και από πολιτική και από οικονομική και εμπορική άποψη. Μας είπατε ότι η Συρία φοβήθηκε ταυτόχρονα μείωση των τελωνιακών εισόδων, αύξηση των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στασιμότητα των δικών της εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ε, βάσιμη όλη αυτή η φόβη της Συρίας ευσταθούν αυτές οι ανησυχίες και υπάρχει τρόπος να διασκεδαστούν αυτές οι ανησυχίες με μια τροποποίηση ενδεχομένω κάποιος παραγράφου της Συμφωνίας Σύνδεσης σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τότε που βγήκε η Συρία από την πολιτική της απομόνωση μετά τη διάσκεψη κορυφής της Ντόχα και τον Ιούλιο του 2008 στη διάσκεψη κορυφής Ευρωμεσογείου υπήρξαν θετικές εξελίξεις και ποιε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο κύριο Σαλαφράγκα. Σας ευχαριστώ. Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις που μας περιέγραψε ο κύριος Μιγκαρέλη και ε, τις εξελίξεις στο Συμβούλιο. Ρωτώ λοιπόν, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή της στάσης του Συμβουλίου και ε, η μετάβαση σε μια πιο θετική στάση η βελτίωση των σχέσεων Λιβάνου-Συρίας ε, ελήφθη υπόψη για να δικαιολογηθεί αυτή η τροπή προ το θετικό στη θέση του Συμβουλίου. Και δεν ξέρω αν ε, είναι φυσιολογικό για το Συμβούλιο ε, να δίνει ένα τελεσίγραφο 10 ημερών, μια διορία στον Υπουργό Εξωτερικών προκειμένου να προσκαλέσει μια χώρα εταίρο για να υπογράψει μια συμφωνία. Για ποιο λόγο ε, δόθηκε αυτή η διορία στον Σύριο Υπουργό από διπλωματική άποψη νομίζω ότι είναι κάπως περίεργος αυτός ο τρόπος δράσης. Επίση, η μονομερή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση που επισύνοψε στη Συμφωνία Σύνδεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι το βασικό στοιχείο που θέλουμε να εισαγάγουμε σε αυτέ τι συμφωνίε σύνδεση δεν τεκμηριώνουν μια πολύ, μια πολύ εφησυχαστική στάση. Ε, και όταν μας μιλήσατε προηγουμένως για την πολιτική κινήτρων και φοβήτρων απέναντι στη Λευκορωσία, όταν μιλούμε για τις μακροοικονομικές δημοσιονομικές ενισχύσεις, υπάρχει το θέμα του δικαιοστασίου του μορατόριου στη θανατική ποινή. Στην περίπτωση Λευκορωσίας το χρησιμοποίησατε αυτό ε, ή και στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη Συρία, το θέμα της, του μορατόριου της θανατικής ποινής είναι πολύ σημαντικό, θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε κύριε κύριος Πέτερινγκ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μιγκαρέλη για το έργο που κάνει σε έναν τομέα τεράστιας σημασίας. Η Συρία είναι μια χώρα κλειδί για τη Μέση Ανατολή. Πρέπει να εκτιμήσουμε την σημασία τους. Ο κύριος Αλαφράνκα ανέφερε ήδη το Λίβανο και θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος του Νίκ Μποντή. Η Συρία είναι σημαντική σχέση με το Ιράν και εάν θέλουμε να χαλαρώσουμε τις σχέσεις Συρίας-Ιράν πρέπει να αποκτήσουμε εμεί ισχυρότερε σχέσεις με τη Συρία και η Συρία μπορεί να συνεισφέρει στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δηλαδή χρειαζόμαστε την Συρία να αναφερθώ τώρα και εγώ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέρσι επισκέφτηκα τη Συρία, μίλησα με διάφορους ηγέτες διαφόρων θρησκειών και νομίζω πως ε, η θρησκευτική ελευθερία υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό από τα περισσότερα αραβικά ε, κράτη και μου είπαν όλοι για τους θρησκειών πως υπάρχει συνεργασία με χριστιανούς και μουσουλμάνους και με τις υπόλοιπες θρησκείες ταυτόχρονα ε, πράγματι εάν υπήρχε μονομερής δήλωση δική μας είναι σωστό αυτό και θέλω να ενθαρρύνω και τον κύριο Σάρκοζη ο οποίος με την Σύνοδο Κορυφής Μεσογείου στις 30 Ιουλίου ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία έτσι ώστε και με τις ε, διμερείς ε, σχέσεις, δηλαδή εμπροκειμένο της Γαλλίας, αλλά και όλοι μαζί από κοινού πρέπει να εμπλακούμε με τη Συρία. Αυτή είναι η δική μου πολιτική σύσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ανησυχώ για το ότι εξακολουθούν στη Δαμασκό να υποστηρίζουν ε, τρομοκρατικά δίκτυα όπως η Χαμάς, Χεσμπολάχ και η Ισλαμική Τζιχά. Τι κάνει η Κομισιόν. Ανησυχώ για το ότι δόθηκε ρωσικό πολεμικό υλικό συγκεκριμένα στη Χεσμπολάχ στις οργανώσεις αυτές και υπάρχει στενή σχέση άξονας θα έλεγα Τεχεράνης Δαμασκού. Επίσης υπήρχε μια μυστηριώδης έκρηξη σε μια βόρειο-κορεατική μάλλον πιστεύουμε ερευνητική εγκατάσταση στη Συρία. Επίσης πιθανώς υπάρχουν χημικά και βιολογικά όπλα. Πιθανότατα κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει για μια σχετική ρήτρα για να ξεφορτωθούν αυτά τα χημικά όπλα. Αλλά τι απέγινε τελικά γιατί δεν το παρακολούθησα και ένα λεπτό ζήτημα. Η έρευνα στην δολοφονία του Χαρίρη υπό τον ΟΗΕ. Τι θα γίνει εάν κατονομαστούν ε, στελέχη της κυβέρνησης ή των μυστικών υπηρεσιών ότι έχουν σχέση με αυτή τη δολοφονία. Θα θέλατε να απαντήσετε κύριε Μιγκαρίλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριο Μπόντι έκανε τρεις ερωτήσεις. Ε, η ειδικότητα της, τη συμφωνία σε σχέση με τη συμφωνία σύνδεση με τους ε, Άραβες ε, γείτονες. η ειδικότητα είναι η δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε όλες τι συμφωνίες αυτού του τύπου πρέπει να πούμε ότι η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικό στοιχείο της συμφωνία Αν ένα από τα μέρη, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση προφανής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σε θέση να αναστείλει την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας ανα πάσα στιγμή. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την μονομερή δήλωση δεν προσθέτει τίποτα είναι θέμα πολιτική βούληση. Γνωρίζω χώρε, δεν θέλω να τι κατονομάσω για να μην δημιουργήσω πρόβλημα, όπου είχαμε τέτοιε συμφωνίε και όπου υπήρχαν παραβιάσει προφανεί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όμω δεν προβήκαμε σε αναστολή. Και δεν μιλάω για χώρε τη περιοχή κατά ανάγκη. Και σε άλλε περιοχέ του πλανήτη είχαμε τέτοια προβλήματα με μεγάλε χώρε. Είναι θέμα πολιτική βούληση. Το Συμβούλιο έχει την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή αυτή τη ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να αναστείλει την εφαρμογή τη συμφωνία. Υπάρχει πάντως αυτή η δίκευση ε, που είναι αυτή η μονομερής δήλωση. Ε, έχουμε αυτή η μονομερή δήλωση γιατί ένα κράτος μέλος ε, μας δημιουργούσε προσκόμματα και για να αρθούν τα προσκόμματα χρειάστηκε να δεχτούμε αυτή τη μονομερή δήλωση. Οι φόβοι των Σύριων είναι βασισμένοι. Τα πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα ποτέ, ούτε εδώ. Είναι σαφές ότι βραχυπρόθεσμα η εφαρμογή μιας τέτοιας συμφωνίας θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιες δυσκολίες σε οικονομικούς ε, τομείς που είναι ευπαθείς. Όταν ανοίγεται μια οικονομία που μέχρι τώρα ήταν να κλειστή στο διεθνή ανταγωνισμό, υπάρχουν τομείς που μέχρι στιγμής προστατευόταν και που δεν είναι αρκετά εξοπλισμένοι για να αντισταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στη Συρία. Ε, αλλά μπορεί να συμβεί και σε οποιαδήποτε οικονομία ανοίγει προς τα έξω, ε, βραχυπρόθεσμα μπορεί να συμβεί αυτό. Ε, βραχυπρόθεσμα λοιπόν θα υπάρξει ε, μείωση των τελωνιακών εσόδων. Παρότι δεν θα είναι στο ύψος αυτών που ισχυρίζονται οι ΣΥΡΙ. Ε, προσπαθήσαμε με κάποια επιχειρήματα να τους εξηγήσουμε ποια θα είναι βραχυπρόθεσμα, οι απώλειες από τα τελωνιακά έσοδα, αλλά μεσοπρόθεσμα και βραχυ, μακροπρόθεσμα τι πρόκειται να κερδίσουν. Ε, πάντως, η, κυβέρνηση της Συρίας, όπως κάθε κυβέρνηση, προσπαθεί να ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού της. Γι' αυτό θα πρέπει να εξυγχρονίσει την οικονομία και επομένως να ανοίξει προοδευτικά προς τα έξω. Αυτή η κίνηση, αυτή η προσπάθεια, η τάση έχει ξεκινήσει. Και εμείς με τη συμφωνία θέλουμε να συνοδεύσουμε αυτή την κίνηση. Επίσης εξηγήσαμε στους Σύριους, φίλους, ότι έχουμε ένα προπολογισμό ε, συνεργασίας που υπομορφή ε, τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βοηθήσουν τις βιομηχανίες τους και, την, και τις επιχειρήσεις τους σε πολλούς τομείς. Ε, επομένως, ε, βραχυπρόθεσμα θα υπάρξουν ενδεχομένως δυσκολίες, αλλά υπάρχουν ε, μέσα για να μειωθούν αυτές οι βραχυπρόθεσμες δυσκολίες, ούτω ώστε να κερδίσει ουσιαστικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η Σύρια. Ε, ίσως είναι λίγο δικολαβίστικη η απάντηση, αλλά δεν μπορώ να σα απαντήσω ναι όχι. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά σταθερή θα έλεγα. Ε, να απαντήσω τον κύριο Σαλανφράγκα ε, γρήγορα. Γιατί αλλάξαμε προσέγγιση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί απλούστατα η Συρία βελτίωσε τις σχέσεις της με πολλούς ε, γειτονέ τη. και κυρίως με το Λίβανο, όπως είπατε κι εσείς. Γνωρίζετε πολύ καλά το Λίβανο και ξέρετε ότι η Συρία για πρώτη φορά έχει διπλωματικές σχέσεις με το Λίβανο. Ε, έχει δημιουργήσει μια πρεσβεία και έχει διορίσει ένα πρέσβη στο Λίβανο. Αυτό είναι σημαντικό βήμα. Υπάρχει μια συνεργασία με άλλες όμορες χώρες. Ξέρετε ότι μέχρι πρότινος η Συρία είχε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, με το Ισραήλ μέσω της Τουρκίας. Σήμερα είναι σε νεκρό σημείο, αλλά τουλάχιστον έγινε μια προσπάθεια. Ε, έγιναν και οι Λιβανέζικες εκλογές που διεξήγησαν καλά. Ε, δημιουργήθηκε μια κυβέρνηση εθνική ενότητα στο Λίβανο. Ε, όλα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα, αλλά μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσαν και χειρότερα. Ε, σε πολλούς τομεί, λοιπόν, η Συρία έπαιξε ένα θετικό ρόλο στην περιοχή και θα πρέπει να το καταγράψουμε αυτό. Τώρα, δέκα μέρες αρκούν για να επιτρέψουμε στον Υπουργό Μουάλαμ να έρθει. Δεν θέλω να υποκαταστήσω τη Σουηδική Προεδρία, αλλά δεν μπορούμε να τους πιέσουμε όταν ε, πέρασαν τέσσερα χρόνια έτσι. Τώρα, τι κάνουμε το Χεσμπορλά και το την Αμάς, ε, ρώτησε ο κύριος Τάνοκ. Όταν συζητάμε με τη Συρία, ε, τους ζητάμε να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους, ούτως ώστε αυτές οι δύο οργανώσεις να παίξουν ένα πιο θετικό ρόλο στη Γάζα και στο Λίβανο. Και κάθε φορά που συζητούμε με τις ε, αρχές της Συρίας αυτό κάνουμε, αυτό ζητάμε. Επίσης προσπαθούμε να σκεφτούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τους Λιβανέζους να ελέγξουν τα σύνορα Λιβάνου-Συρίας. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουν ένα μεγάλο τμήμα του εξοπλισμού της Χεσμπολά περνά από αυτά τα σύνορα. Επομένως, ε, έχουμε διάλογο με τις Συριακές Αρχές για να τους εξηγήσουμε ότι μια και έχουν επιρροή σε αυτές τις διοργανώσεις, θα ήταν ευκταίο να ασκήσουν μία έτσι, επιρροή, ούτως ώστε να είναι, γίνουν πιο μετριοπαθείς, αν θέλετε, αυτές οι οργανώσεις. Τώρα, όπλα μαζικής καταστροφής. Υπάρχει στη συμφωνία μία ρήτρα μέσω της οποίας τα δύο μέρη, η Σύρια προκειμένου, ε, δεσμεύεται να καταπολεμήσει την εξάπλωση των ε, όπλων μαζική καταστροφή. Φυσικά θα πρέπει να εφαρμοστεί και θα πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση να ελέγξουμε την εφαρμογή αυτή τη ρήτρα. Τώρα, η δολοφονία του ε, Πρωθυπουργού Χαρίρη. Δεν ξέρω τι θα ανακαλύψει το δικαστήριο, δεν θέλω να προδικάσω τα απορίσματα του δικαστηρίου. Η Κομισιόν πάντως χρηματοδοτεί το δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη λειτουργία αυτού του δικαστηρίου, ούτως ώστε να, δοθ, να χυθεί άπλετο φως στις πολιτικές δολοφονίες του Λιβάνου και κυρίως τη δολοφονία του Πρωθυπουργού κ. Χαρίρη. Τελευταίο θέμα νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Και είναι μια προκαταρτική συζήτηση. Προσοχή, έτσι δεν υπάρχει βασικό κείμενο, το λέω. Είναι προκαταρτική συζήτηση. Και είναι μια ευκαιρία για τους συναδέλφους να απευθύνουν στον εισηγητή τις απόψεις τους. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Αρλάκη. Σας ευχαριστώ, Η πρόθεσή μου με την έκθεση... Δεν είναι να επαναλάβω άλλα έγγραφα ή άλλες ε, στρατηγικές. Θα ήθελα δύο λεπτάκια να μιλήσω για το προφίλ της έκθεσης και μετά να ζητήσω από τους συναδέλφους προτάσεις. Το πρώτο στοιχείο της έκθεσης είναι η συνολικότητα χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα είναι έτσι μια γενική έκθεση που θα παραβλέψει τα εμπειρικά δεδομένα και τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Θέλω λοιπόν τις απόψεις σας για τρεις τομείς ε, που μας ανησυχούν και πρέπει να ερευνηθούν πρώτα απ' όλα. Να δούμε τι έχει γίνει ήδη από πλευράς στρατηγικής για το Αφγανιστάν τα τελευταία 8 χρόνια. Μετά την παρέμβαση του Οκτωβρίου 2001. Να μετρήσουμε τον αντίκτυπο της ξένης μη στρατιωτικής παρέμβασης ειδικά όσον αφορά την βοήθεια στην χώρα από τις μεγάλες χώρες, δηλαδή η η Ιαπωνία και την Ευρώπη και άλλες χώρες. Θα προσπαθήσω να κάνω μια αξιολόγηση των τομέων της προηγούμενης έκθεσης, δηλαδή που είχαμε, αντίκτυπο που δεν είχαμε. Είναι σαφές πως χρειάζεται να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά γιατί ο αντίκτυπος αυτός είναι επαρκής Σήμερα το πρωί ο Αφγανός πρέσβης της Βρυξέλλες ήρθε στην ε, αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν και μας παρουσίασε την κατάσταση της διεθνούς βοήθειας από τη σκοπιά της Αφγανιστής, αυγανικής κυβέρνησης και του αυγανικού λαού που είναι πολύ ανησυχητική η εικόνα αυτή. Θα ήθελα λοιπόν στην έκθεση να αφιερώσουμε και λίγο χώρο στην άποψη αυτή, όχι μόνο στην άποψη των δωρητών και της διεθνούς κοινότητας, αλλά και στην άποψη και την οπτική των αυγανών και των αυγανικών αρχών. Δεν τους ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται η διεθνής βοήθεια. Παραδέχτηκε ο κύριος Πρέσβης τη μεγάλη διαφθορά και, την κατασπατάληση της βοήθειας, αλλά ανέφερε και ένα πρόβλημα που θα ήθελα και εγώ να αναφέρω, πως υπάρχει στην αλυσίδα αυτή της βοήθειας κατασπατάληση και διαφθορά δίνουμε γύρω στο 1 δισεκατομμύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για μια τεράστια, τεράστιο ποσό. Μιλάμε δηλαδή για μια χώρα που έχει 10 δισεκατομμύρια ΕΠ και εμείς τους δίνουμε 1 δισεκατομμύριο. και πρέπει να δούμε πώς δίνεται αυτή η βοήθεια και ποιος είναι ο αντίκτυπος. Και επί τη ευκαιρία, με την, επί τη ευκαιρία της έκθεσης να δούμε τι γίνεται με την καλλιέργεια της Παπαρούνας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ε, γιατί αυτό έχει σημασία για εμάς. Ε, είναι πηγή του 95% της ηρωίνης και της μορφίνης και των οπιούχων που καταναλώνονται στην Ευρώπη. Και θα προσπαθήσω επιτέλους να μπει σοβαρά αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Γενικές αναφορές στο εθνικό σχέδιο του Αφγανιστάν ε, κατά πολέμηση των ναρκωτικών δεν αρκούν. Θα ήθελα, αν συμφωνείτε, να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα. Στην καταπολέμηση της καλλιέργειας Παπαρούνας έχω συγκεκριμένη εμπειρία όταν ήμουν εκτελεστικός διευθυντής ε, Τη Υπηρεσία καταβολή των Ναρκωτικών, το ΟΗΕ, είχα μια σχετική πρωτοβουλία, μιλάμε για πριν από μια δεκαετία. Τα οικονομικά μέσα, οι πόροι ε, σήμερα είναι τεράστιοι σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, οπότε πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά. Τέλος, η εκπαίδευση της ε, Αφγανικής αστυνομίας. Όπως ξέρετε κάθε νέα στρατηγική ε, για το Αφγανιστάν από τις ε, από τις ΗΠΑ την Ευρώπη έχουν ως ε, βασική πτυχή την εκπαίδευση της αστυνομίας του Αφγανιστάν για να αναλάβουν κάποτε και μάθαμε σήμερα πως ο πρόεδρος Ομπάμα θα θέσει χρονοδιαγράμματα Πολύ σημαντικό αυτό για όλους όσου ασχολούνται με μια μη στρατιωτική στρατηγική για το Αφγανιστάν. Θα σταματήσω εδώ για την εκπαίδευση της αστυνομίας. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Αλλά βεβαίω είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Il primo intervento è quello richiesto dal collega Thaler. Ο Στάλιν είναι ο πρώτος ομιλητής. Thank Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, νομίζω πως ε, η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρωτοβουλία που ενέλαβε. Είναι σημαντική γιατί αφενός ε, μας δίνει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρούμε την εξωτερική μας πολιτική και την πολιτική ασφαλεία Οχτώ χρόνια ακολουθούμε την Ουάσιγκτον. Την Ουάσιγκτον. Αυτοί είχαν τους λόγους τους. Μπήκαν εκεί το 2001, πέρασαν 8 χρόνια, και αποτέλεσμα 0. 8 χρόνια δεν κράτησε ούτε ο δεύτερος παγκόσμιος. Και το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι μήνα με το μήνα ο αριθμός των Ταλιμπάν αυξάνεται. Όσο περισσότερους στρατιώτες στέλνουν οι συμμαχικές δυνάμεις, τόσο περισσότερου Ταλιμπάν δημιουργούμε. Είναι απαράδοξο. παράδοξο. Η στρατηγική αυτή δεν έχει επιτύχει. Πρέπει να βρούμε μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Ο τίτλος σας. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται μια λογική προσέγγιση και μια έξυπνη λύση για να αποσυρθούμε από το Αφγανιστάν. Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε οτιδήποτε δεν εμπίπτει στην κατηγορία Ταλιμπάν να το ενθαρρύνουμε. Όσους δεν είναι ακραίους να υπάρξει αυτοδιοίκηση, να αρχίσουν να κυβερνούν τη χώρα μόνοι τους. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει τη στρατηγική της και να την ακολουθήσει ανεξαρτήτως του πόσο χρειάζονται οι Αμερικάνοι για να καταλάβουν ότι αυτός ο πόλεμος δεν κερδίζεται. Ένα δυσάρεστο έργο. Θα πρέπει να σας ανακοινώσω ότι σε 10 λεπτά οι διερμηνείς αποχωρούν. Και έχουμε ακόμα 7 ομιλητές. Θα ήθελα να ακούσουμε όλους τους ομιλητές, αλλά ζητώ από όλους να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα. Ο κύριος Αλαφράγκα είναι ο πρώτος. Με αυτό το πνεύμα παρακαλώ όμω να παρέμβετε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση. Το πρόβλημα αυτό του Αφγανιστάν θα πρέπει να το εστιάσουμε με σφαιρικό τρόπο. Γιατί έχουμε τον αντιτρομοκρατικό αγώνα και τον αγώνα κατά της εξέγερση, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την υποχρέωση να σταθεροποιήσουμε τη χώρα. Ο πρόεδρος Ομπάμα άργησε τρεις μήνες για να υιοθετήσει μία έκθεση μετά την απεσιόδοξη έκθεση που το έκανε ο διοικητής Μακρίσταλ τον ε, ο, αρχηγός των επιχειρήσεων και έδωσε μία πολύ αρνητική εντύπωση για τις δυνάμεις του ΑΙΣΑΦ σε ό,τι αφορά την προστασία του αυγανικού πληθυσμού. Γιατί ο αφγανικός πληθυσμός εκλαμβάνει τον ΑΙΣΑΦ ως ε, δύναμη εισβολής παρά δύναμη προστασίας. Τα στοιχεία που μας δώσατε για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εντυπωσιακά. Με αυτή την άποψη πάντως η εικόνα που δίνει και οι σύμμαχες δυνάμεις της ΑΙΣΑΦ αλλά και οι δυνάμεις της, ε, των ΗΠΑ ε, δείχνουν πενιχρά αποτελέσματα που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος των τεράστιων πόρων που διαθέτει η διεθνής κοινότητα στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρό τρόπο λύσεις ε, που θα επιλύσουν αυτή την πολύ σοβαρή πρόκληση, θα αναλάβουν αυτή την πολύ σοβαρή πρόκληση που έχουμε στο Αφγανιστάν. Ο κύριος Κουαλτιέρη. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ενδιαφέρουσα εισαγωγή του, που μπορώ να την ε, συμμεριστώ καταρχήν. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του Αφγανιστάν, πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη διπλή αντίφαση που ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Αφγανιστάν. Από τη μία, οι πόροι που διοχετεύονται ε, προς το Αφγανιστάν είναι πάρα πολλοί και από την άλλη πρέπει να ε, συμμετάσχει και στις συμμαχικές επιχειρήσεις. Η δεύτερη αντίφαση. Υπάρχει το θέμα του comprehensive approach για το Μαρλακάντ. Από την άλλη, όμως, δίνεται έμφαση στην αύξηση των στρατιωτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει απτά, απτές χειρονομίες, χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα. Φυσικά, η δέσμευση των, των ΗΠΑ είναι πολύ σημαντικό σημαντική και η στρατηγική που ξεκίνησε ο πρόεδρος Ομπάμα θα καθορίσει τις εξελίξεις τους επόμενους μήνες. Αλλά υπάρχει και χώρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεισφέρει και εκείνη ε, και να διαμορφώσει τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσει ε, στις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το action plan είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει ε, να υπάρξουν περισσότερα σε επίπεδο συνέπειας και συνεκτικότητας. Γι' αυτό θα ήθελα ο εισηγητής να ε, εξετάσει τις αποστολές της ΚΕΠΑ, ΕΠΑ, και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα διευρύνει την αποστολή της και στον τομέα της δικαιοσύνης. Ο κ. Γκζίμπ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προτινόμενη στρατηγική για το Αφγανιστάν και την τοποθέτησή του. Καταρχήν ε, υπήρξε μια απογοήτευση με το θέμα, με την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Παρόλο που ε, γίνεται έκκληση προς συμμάχους να αυξήσουν τη στρατιωτική του παρουσία εκεί και αρχίζει η δεύτερη θητεία του Πρόεδρου Καρζάη που ε, ζήτησε συγγνώμη από, το, από τους Ταλιμπάν για την κατοχή των εδαφών και τις απειλές κατά της ειρήνης. Δεν θα μπορούσαμε στην έκθεση αυτή να αναφερθούμε σε αυτή την παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και τι μέσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε ένα τμήμα αυτών που δίνουν μάχη κατά των, της παρουσίας μας να συμμετέχουν στην συνεργασία. Επίσης, ε, ε, έγιναν δηλώσει ότι το Αφγανιστάν απομακρύνεται από την αλκαΐδα και από τις ε, με την τρομοκρατία. Ο κύριος Λέζινγκ, η κυρία Λέζινγκ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να αναφερθώ σε μια πτυχή που αναφέρθηκε και πρέπει να δούμε κάπως πιο προσεκτικά στην έκθεση το κόστος. Έχουμε 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια που προτείνονται για τον στρατό και την αστυνομία και έχουμε 890 εκατομμύρια που είναι ο προϋπολογισμός στο Αφγανιστάν. Πώς πάει η ε, κατάσταση. Δηλαδή αν αποσυρθούμε θα έχουμε ένα στρατό και μια αστυνομία που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί κάπως. Ε, αυτοί θα πέσουν πάνω στον πληθυσμό και θα τον φάνε. Πρέπει να το σκεφτούμε να έχουμε πολύ συγκεκριμένες ιδέες για το τι θα γίνει στο μέλλον και μετά συγκεκριμένα ερωτήματα. Πόσοι υπάλληλοι της Ένωσης βρίσκονται εκεί στο πλαίσιο της EU pol Πότε θα φτάσουμε το όριο των 500 ε, όσον αφορά αυτή την δύναμη και όπως ζητάει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και πώς έχει συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και μετά για την αστυνομία ισχύει πως ε, θα αποσταλούν 500 ε, άνδρες της ευρωπαϊκής δύναμης ε, από του χρόνου και ποια θα είναι η συνεργασία με την εκπαιδευτική δύναμη του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Βάγγελ. Ευχαριστώ. Ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν τράβηξε πολλά χρόνια. Και έχουμε εκεί έμπειρους ανθρώπους με στρατιωτική πείρα, με στρα... πείρα στα ανθρωπιστικά και στα πολιτικά θέματα. Και αντί να ακούμε και να εκμεταλλευόμαστε την πείρα αυτών των ανθρώπων, έχουμε όλο και νέα σχέδια για αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας, κάτι που προϊονίζεται συνέχιση του πολέμου. Στον πόλεμο αυτό δεν θα υπάρξει κανένας νικητής, μόνο χαμένοι. Και έτσι αντιλαμβάνομαι την τελευταία δήλωση περιτακτικής του Προέδρου Ομπάμα. Κατά τη γνώμη μου, η τελευταία αναγγελία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική και δεν μας δημιουργεί καμία διάθεση αισιοδοξία και χαράς. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία που ανέλαβε στην έκθεση του κύριο Σαρλάκη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα επιπλέον στοιχείο. Αναφέρθηκε από τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών χθε ότι το Αφγανιστάν ουδέποτε δεν είχε στην ιστορία του μια κεντρική κυβέρνηση. Και τώρα θέλουμε μια χώρα με κεντρική κυβέρνηση. Ενώ ο Αφγανικό λαό είναι κατά μια τέτοια κεντρική κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται καν μια τέτοια κεντρική κυβέρνηση γιατί αντιβαίνει στι παραδόσει του. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή μας, τον κύριο Αρλάκη, για την ε, θέση που υιοθέτησε. Τελευταίες παρεμβάσει του κυρίου Τάνοκ και του κυρίου Νίλσεν. Σύντομα. Καλή τύχη κύριε Αρλάκη. Ελπίζω Νομίζω πως η πρώτη φράση τα λέει όλα. Το να γυρίσει σελίδα το Αφγανιστάν και το Πακιστάν είναι φοβερή πρόκληση. Ε, τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά. Θυμάμαι που είχαμε αυτή τη συζήτηση το 2001-2002. Και τίποτα δεν έχει αλλάξει παρά το ότι πλέον υπάρχει αυτή η έννοια του ΑΦΠΑΚ εδώ πέρα, Αφγανο-Πακιστάν ένα σημαντικό ζήτημα που υπάρχουν Ταλιμπάν και στις δύο πλευρές των συνόρων και αποσταθεροποίηση δηλαδή του Πακιστάν και βεβαίως το ότι η κυβέρνηση του Πακιστάν ακόμα δεν έχει αποφασίσει να εξαλείψει τους τζιχαντιστές στο έδαφος της. Επίσης η βοήθεια, η στρατιωτική που τους δίνουμε τόσο καιρό δεν πάει για να καταπολεμήσει την ε, εξέγερση, απλά μιλάμε για στρατιωτικό εξοπλισμό στα σύνορα του, του Πακιστάν και δεν έχουν καταφέρει να τους νικήσουν τους Ταλιμπάν στο το Είναι σοβαρά αυτά τα ζητήματα, συμφωνώ μαζί σας πως ε, το εμπόριο των ναρκωτικών είναι μεγάλο. Ε, πριν από 5 ή 6 χρόνια, έτσι, ηρωνικά ως ε, γιατρός, είχα πει πως θα έπρεπε να συλλέξουμε όλες τις παπαρούνες και να τις κάψουμε και να τους πληρώσουμε μετρητά. Είναι λιγότερα από τα 3,5 δισεκατομμύρια που στέλνουμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στρατεύματα βεβαίως, αλλά είναι πράγματα κατόρθωτα. Ευχαριστούμε. Κύριε Τάνοκ, παρακαλώ. Φυσικά θα πρέπει να ξεφύγουμε από την αυγανική παγίδα στην οποία μας εγκλώβησε ο George Bush. Πότε? Αυτό θα το κρίνουμε προσδιορίζοντας ένα χρονοδιάγραμμα από κοινού με τους Αφγανούς και φυσικά αναμειγνύοντας και την ευάλωτη και νέα κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν που υπάρχει όμως και κυρίως τις γυναικείες οργανώσεις του Αφγανιστάν. Είναι αδύνατο να, να πετύχουμε οτιδήποτε χωρίς διαβουλεύσει μαζί τους. Σε ό,τι αφορά την έκθεση Αρλάκη έχω κάποιες παρατηρήσεις. Φυσικά θα πρέπει να ασχοληθούμε με την παρακολούθηση της ε, βοήθειας. Γιατί, γιατί η χώρα αυτή, το, το βυτικό επίπεδο, τρόπο ζωής των δυτικών ε, είναι προσβολή σε μια χώρα που ο πληθυσμός δυναπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης το θέμα της ε, υποστήριξης των Αφγανών ναρκωμανών, γιατί πολλοί Αφγανοί είναι ναρκωμανείς, είναι θύματα των ναρκωτικών, είναι καταναλωτές, χρήστες ναρκωτικών και χρήζουν φροντίδας, περίθαλψης και υποστήριξης. Ό,τι αφορά την αστυνομία, οι μισθοί των αστυνομικών χρειάζονται πολύ πιο υψηλή μισθή για να εξασφαλιστεί μια σοβαρή ε, αυγανική αστυνομία που δεν θα ενδίδει στον πειρασμό της δωροδοκίας τέλος, κάτι που είχα πει και στην συνεδρίαση της αντιπροσωπείας για το Αφγανιστάν, πιστεύω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μια γυναίκα που διοικεί μια περιοχή, την ε, επαρχία του Μπαμιάν στο Αφγανιστάν. Είναι μια καταπληκτική γυναίκα και είναι η πρώτη φορά που μια γυναίκα ε, διοικεί μια περιοχή στην ιστορία του Αφγανιστάν. Και πιστεύω ότι με αυτή τη γυναίκα θα πρέπει να συνεργαστούμε την ε, διοικήτρια της περιοχής του Μπαμιάν. Μπορείτε να σημειώσετε αυτές τις παρατηρήσεις και θα, προβλέψουμε και ένα χρονοδιάγραμμα για μια επόμενη ε, συνάντηση. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν. Ευχαριστώ. Αύριο στις 9 η ώρα, εδώ. No. No, Έχουμε ψηφοφορία αύριο. Εντάξει.